Good morning, colleagues. I know um, some colleagues are pressed for time, so we can make a, a quick start if uh, colleagues would like to take their seats. Thank you. ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ πολύ. Good morning, colleagues. Um, if there are no objections. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Εγκρίνουμε τη μερίσια διάταξη αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις. Δεν έχουμε λετωνικά και δεν έχουμε κροατικά και μαλτέζικα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Ας περάσουμε στην κοινή συζήτηση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις θεωρήσεις έχουμε δύο εισηγητές για το ζήτημα αυτό, τον Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγκουιλάρα, καθώς επίσης και τον κύριο Μπρίς ε, Οχτεφέ. Δεν ξέρω αν... Μάλλον. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις θεωρήσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα δύο έγγραφα εργασία τα οποία έχουν προετοιμάσει δύο μα εισηγητέ. Θα δώσω και στου δύο εισηγητέ το λόγο και στη συνέχεια θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με του υπόλοιπου συναδέλφου, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση και προφανώ μπορεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ξέρω ότι ο κύριο Ορτεφέ πρέπει να αποχωρήσει για να πάει σε κάποια άλλη συνεδρίαση. Ενδεχομένω λοιπόν θα μπορούσαμε να ακούσουμε πρώτα την εισήγηση του κυρίου Οχτεφέ, καθότι τον πιέζει ιδιαίτερα ο χρόνος. Λοιπόν, κύριε Οχτεφέ, μπορείτε να πάρετε πρώτο το λόγο και συνέχεια θα πάρει το λόγο κύριο Σαγκουιλάρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να χαιρετήσω την εξαιρετική συνεργασία που καταφέραμε να είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και με τους σκιώδεις ηγετές ε, όσον αφορά το ζήτημα της θεώρησης περιοδίας ε, και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας στο ίδιο θετικό πνεύμα. Έχετε μπροστά σας ένα έγγραφο εργασίας στα πλαίσια του οποίου προσπάθησα να δώσω κάποιε διευκρινήσει. Καταρχά, ποιο είναι το πλαίσιο τη πρόταση αυτή. Εκ πρώτη όψεω, η δημιουργία αυτή τη νέα θεώρηση, τη θεώρηση περιοδία δηλαδή, προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών και αυτό διότι από ό,τι φαίνεται μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη για το σύνολο του χώρου Σέγγεν μέσω της αύξησης της ε, χρησιμοποίησης της θεώρησης αυτής για τον τουριστικό τομέα. Προσπάθησα λοιπόν να δούμε ποιες απαντήσεις, ποιες πιο συγκεκριμένες απαντήσεις θα μπορούσε να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν ένα νέο μέσο, μία νέα θεώρηση, και συνεπώς ως συνομοθέτες θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά όλες αυτές τις νέες πτυχές του νέου αυτού μέσου και θα πρέπει να αποφύγουμε να δημιουργηθεί ένα μέσο το οποίο τελικά δεν θα είναι αποτελεσματικό. Δεν θα καταφέρουμε δηλαδή να οδηγηθούμε σε μια πολιτική θεωρήσεων η οποία θα είναι αποτελεσματική και αποδοτική. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια που είναι απαραίτητη για το χώρο Σέγγεν και το οικονομικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε δηλαδή να εξισορροπήσουμε τα δύο αυτά συμφέροντα, τους δύο αυτούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μηχανισμό που θα απλούστευε θα καθιστούσε πιο αρμονική τη λειτουργία των κοινοτικών θεωρήσεων και ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να γίνει εύκολα αποδεκτό επίσης από τις προξενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κάποια περισσότερα στοιχεία. Έχω τονίσει εγώ καταρχάς κάποια ζητήματα, η επιλογή της νομικής βάσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εγγραφό, στο μα της μας λέει ότι καλύπτει ένα νομικό κενό μέσω του άρθρου αυτού και ότι βασιζόμενοι στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δημιουργήσει μία θεώρηση περιοδίας που θα επιτρέπει για δύο χρόνια στον δικαιούχο να χρησιμοποιήσει τη θεώρηση αυτή και ουσιαστικά αποτελεί μία σώρευση θεωρήσεων βραχίας διάρκειας. Τώρα, μπορούμε να πούμε όμως ότι το χρονικό διάστημα του ενός ή των δύο ετών που προβλέπεται από το νέο αυτό μηχανισμό συνάδει με την έννοια της σύντομης χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στη συνθήκη. Πρώτο ερώτημα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Οι διάφορες κατηγορίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η πρόταση αυτή θα εξυπηρετήσει περίπου 60 με 120.000 άτομα, αλλά θα μπορούσε να απευθυνθεί και στους πάντες, δηλαδή καλλιτέχνες, ερευνητές, φοιτητές και γενικότερα τουρίστες. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει περισσότερο ποιο είναι τελικά το προφίλ των 60.000 ή 120.000 ανθρώπων που θα αποφεληθούν από την νέα αυτή θεώρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός και είχαμε 500 εκατομμύρια τουρίστες το 2014. Από το Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού έχουν έρθει τα στοιχεία αυτά. Αναφερόμαστε λοιπόν στους ε, τουρίστες που είναι μια πολύ γενική και ασαφής ε, κατεμέ κατηγορία. Ενδεχομένως ε, θα μπορούσαμε να είχαμε και πολύ περισσότερους ετούντες που θα υπερβούν τον αριθμό των 120.000 που προβλέπονται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θέλει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει και κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις όσον αφορά τον αριθμό των δικαιούχων της νέας αυτής θεώρησης και μάλιστα ανακατηγορία, για παράδειγμα φοιτητές, ερευνητές, τουρίστες το καθεξής. Πέρα λοιπόν από το ζήτημα της νομικής βάσης, πέρα από το ζήτημα των 60.000, 120.000 και διαφορετικών κατηγοριών δικαιούχων, έχουμε και το ζήτημα της ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά παρακάμπτει το ζήτημα αυτό, χρησιμοποιεί δύο επιχειρήματα. Λέει καταρχάς ότι τα κριτήρια είναι αρκετά αυστηρά ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των ετούντων και το δεύτερο επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι οι υπήκοοι οι οποίοι δεν υπάγονται πλέον στην υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων προέρχονται ούτως ή άλλως από χώρες οι οποίες είναι ασφαλείς αλλά θα μπορούσε να πει κανεί ακόμα και για χώρε που έχουν υψηλό επίπεδο ασφάλεια όπω η Γαλλία, ότι παρόλα αυτά έχουμε ένα μεγάλο αριθμό παρανόμων μεταναστών ή εγκληματιών που θα μπορούσαν να θελήσουν να χρησιμοποιήσουν ε, ένα τέτοιο νέο μηχανισμό, μια τέτοια θεώρηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση το επίπεδο ασφάλειας να διατηρηθεί πάρα πολύ ψηλό και αυτό θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο προξενείων. Ξέρετε ότι οι εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, έχουν τεράστιες ικανότητες προσαρμογής, μπορούν λοιπόν να βρουν όλα τα κενά του συστήματος και να το εκμεταλλευτούν. Το ζήτημα λοιπόν της ασφάλειας πρέπει να μας απασχολήσει ως τρίτο σημείο και ως τέταρτο σημείο οικονομική ανάπτυξη, οικονομικές επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι θα μπορούσαμε να διηγηθούμε σε επιπλέον έσοδα 500 εκατομμύρια ως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε τήσια βάση, επιπλέον έσοδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία όμω αυτά τα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασιζόμενη σε μελέτες του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εργοδοτικών Ενώσεων στον τομέα των παραστατικών τεχνών. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μία νέα θεώρηση μια θεώρηση περιοδίας. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να αυξήσουμε την οικονομική ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά στα δεδομένα που μας δίνει ένας και μόνος σύλλογος, ο οποίος άλλωστε έχει συμφέρον να δημιουργηθεί αυτή η νέα θεώρηση περιοδίας. Να σας δώσω και κάποια παραδείγματα. Στην Ιαπωνία ένας Γερμανός υπήκος μπορεί να μείνει έξι μήνες χωρίς θεώρηση και ένα Γάλλος τρει μήνες χάρη στις ε, συμφωνίες που ισχύουν αυτή τη στιγμή, χάρη στις τρέχουσες συμφωνίες. Δεύτερο παράδειγμα, ένας Βέλγος, Ισπανός ή Γάλλος, υπήκος οποιοδήποτε άλλη χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται να έχετε θεώρηση προκειμένου να μείνετε να περάσετε από τον Καναδά. Η γαλλος υπηκος οποιοδηποτε αλλης χωρας ευρωπαικης ενωσης δεν Επιτροπή ζητά τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν διμερεί συμφωνίες με τις τρίτες χώρες να προβλέψουν μία αρχική μεταβατική περίοδο πέντε ετών. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη όμως τα ζητήματα αμοιβαιότητος όσον αφορά τις διμερείς αυτές συμφωνίες. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένως και το Συμβούλιο, θα ήταν σε θέση να μας δώσουν ένα κατάλογο όλων αυτών των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Δεν έχουμε ακόμα αυτόν τον κατάλογο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διασυνδέσει το νέο αυτό σύστημα, προβλέπει τη νέα αυτή θεώρηση περιοδίας, με το νέο σύστημα εισόδου και εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ε, η πρόταση ε, απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών ετούντων από την υποχρέωση λήψη ακτιλικών αποτιμάτων ενδεχομένω να μην λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται πάντα στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση η λήψη δακτυλικών αποτιμάτων. Επίση, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση αντικτύπωση όσον αφορά τη νέα αυτή πρόταση θεώρηση ε, περιοδία. Θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να καταγράψουμε τον ενδεχόμενο οικονομικό αντίκτυπο της ε, θεώρησης αυτής, αλλά να δούμε επίσης και ποιο θα είναι το διοικητικό άχθος, ιδίως για τις προξενικές αρχές στις χώρες εκείνες, οι οποίες θα επιβαρυνθούν περισσότερο λόγω της διεκπαιρέωσης αυτής της νέας θεώρησης περιοδίας. Πρέπει επίσης να δούμε και ποια θα είναι η θέση των τρίτων εκείνων χωρών που έχουν διμερείς συμφωνίες με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τελικά η νέα αυτή θεώρηση περιοδίας θα λειτουργήσει θετικά, ελκυστικά ή αποτρεπτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία όσον αφορά την οικονομία, την ασφάλεια της νέας αυτής θεώρησης και Έχουμε μια νέα πολιτική όσον αφορά τις θεωρήσεις, μια κοινοτική πολιτική η οποία λειτουργεί θετικά. Έχουμε το χώρο Σέγγεν που είναι ένας καταπληκτικός χώρος κινητικότητας αλλά που έχει και αυτό τα όρια του γιατί έχουμε δει ότι πολλές φορές υπάρχει διασυνοριακή μετακίνηση κλιματικών ομάδων και μολονότι πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την νέα αυτή πρόταση, καθότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε ότι η νέα αυτή θεώρηση σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει αντικείμενο κατάχρηση και επίση θα πρέπει να είναι αρκετά ελκυστική προκειμένου πραγματικά να οδηγήσει σε περισσότερο πλούτο, σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση clear Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε θέσει πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριο Λόπες Αγιλάρο, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την εκτιμησή μου προς το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί και το οποίο μόλις μας εξέθεσε ο κύριος Οχτεφέ. Εδώ και μήνες έχουμε συνεργαστεί, είχαμε συναντήσεις και το έγγραφο εργασίας το οποίο αποβλήθηκε συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσω σήμερα στο πρώτο αυτό σημείο της ημερήσιας διάταξης επιτροπής μας. Το δικό μου έγγραφο αφορά ε, την αναδιατύπωση του λεγόμενου κώδικα των θεωρήσεων. Και τα δύο αυτά θέματα θα πρέπει να εννοηθούν ε, και να γίνουν αντιπτά ως ένα πακέτο και η αναδιατύπωση του κώδικα θεωρήσεων και η πρόταση του κυρίου Ορτεφέ για μια θεώρηση περιοδία. Συνδέονται τα δύο αυτά θέματα και έχει στη σημασία να καταλάβουμε ότι εάν τα χειριστούμε και τα δύο θέματα παράλληλα, θα είναι ιδέωσα διαδικασία. Εάν μας διαφύγει η διασύνδεση των δύο ζητημάτων, ίσως ε, αντιμετωπίσουν προβλήματα που δεν τα περιμέναμε. Share the, uh, the uh, explanation of... Συμφωνώ με τους στόχους, όπως μας τους εξέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο κύριος Ορτεφέ εξήγησε και αυτός ακόμη περισσότερο τα σχετικά ζητήματα 90 ημέρες μέσα σε 180 ημέρες μπορεί να μείνει κάποιος που έχει αυτή τη θεώρηση αρκεί να μην μείνει πάνω από 90 ημέρες στο ίδιο κράτος μέλος. Πολύ χρήσιμο εργαλείο για καλλιτέχνες, για παράδειγμα, για αθλητές, για ερευνητέ. Ιδίω άμα μιλάμε για ανταλλαγές πολιτιστικές, επιστημονικές. Γενικώ έχουμε μεγάλη κινητικότητα επαγγελματιών και αυτό θα διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική τύπου για την καταλληλότητα αυτής της θεώρησης περιοδίας. Καταλαβαίνω και κατανοώ τις ανησυχίες της και τα επιχείρηματά του. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι όσοι νομοθέτες, από κοινού δηλαδή με το Συμβούλιο, πάντα βάση πρωτοβουλία της Κομισιόν, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό να μην παρεμποδίσουμε την ορατότητα, την προβολή Ε, και την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής που πρέπει όπως είπα να γίνει από κοινού κώδικας θεωρήσεων και θέμα ορτεφέ. Η μελέτη αντικτύπου θα μπορούσε να καθυστερήσει την έγκριση της θεώρησης περιοδίας. Άρα και αναδιατυπωμένη εκδοχή του κώδικα θεωρήσεων θα καθυστερούσε και δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Η Θεώρηση περιοδίας, ναι, πράγματι είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σημαντική για αυτό το πεδίο πολιτικής. Αναφέρονται και κάποια αριθμητικά στοιχεία στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προβλέπει ότι από αυτές τις θεωρήσεις θα μπορούσαμε να έχουμε από 500 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως ε, ως ε, κέρδη ε, από την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και πολιτισμικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, επιστημονικές συναλλαγές σίγουρα θα βελτιωθούν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να, να κολλησιεργήσουμε και ούτε θα πρέπει να μείνουμε στη διάρκεια παραμονής. Πρέπει να δούμε και βέβαια και τις επιπτώσεις που θα είχε. Η ολοκλήρωση και των δύο πρωτοβουλειών. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος Σορτεφέ. Όμως, αυτό το οποίο εγώ αποσκοπώ είναι να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, τις ανεπάρκειες αδυναμίες που μας εξέφερε ο κύριος στην ε, παρουσίασή του μόλις πριν και συνεχίζοντας τη συνεργασία μας και κινούμενη παράλληλα ελπίζω να μπορέσουμε να προωθήσουμε την έγκρισή του πακέτου. Δηλαδή, συμπληρωματικά προς το θέμα το πολύ σημαντικό της αναδιατύπωσης κωδικαθήρισεων, να προχωρήσει και το θέμα της αγορήσης περιοδίας. Ευχαριστώ πρόεδρος, ο κύριος ε, Ντεπρέν, ο πρώτος ομιλητής από τους βουλευτές ομάδας μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της, αλλά και για την καλή της διάθεση απέναντι και στον εισηγητή, στους εισηγητές, αλλά και στους υπόλοιπους βουλευτές, γιατί μας παρουσίασε πάρα πολύ διεξοδικά το περιεχόμενο των προτασιών για να μπορούμε και εμείς να εκφράσουμε τις απόψεις μας και ενδεχομένως τις ενστάσεις μας. Εμείς συμφωνούμε ως ομάδα με τον επιδιωκόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχο, δηλαδή ε, να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση ε, τρίτων ε, ε, χωρών, καλόπιστων βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, στο χώρο Σέγγεν. Δηλαδή δεν θέλουμε στον πρώτο τυχόντα και κυρίως σε ταραξίες ε, οι άτομα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ασφάλεια να εισέλχονται πιο εύκολα στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Σε ό,τι αφορά τα ε, προσδοκόμενα κέρδη ιδίω από την ε, θεώρηση περιοδίας, εγώ είμαι πιο επιφυλακτικός. Είμαι χρόνια Ευρωβουλευτή και αν προσθέσω τι θέσει εργασία που θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί από όλε τι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε ένα άνεργο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην πω ότι θα έπρεπε να είχαμε προσλάβει εκατομμύρια επικόστριτων χωρών. Θα μπορούσα να σα δώσω και λεπτομέρειε. Βλέπουμε λοιπόν από την σημερινή κατάσταση ότι πολλές φορές ε, προσκρούει στην πραγματικότητα και στους περιορισμούς της ε, η εκτίμηση της Επιτροπής σε σχέση με ορισμένα αριθμητικά στοιχεία. Έρχομαι τώρα στην ουσία και ξεκινώ με τη θεώρηση περιοδίας. Πρώτα απ' όλα, τα θέματα που θέτει ο κ. Σορτέφ είναι θεμητά. Ε, αναφέρομαι και στην νομική βάση, στην ανάγκη του μηχανισμού, σε αυτά τα 500 εκατομμύρια άτομα που έρχονται κάθε χρόνο στην Ένωση, 60 με 120.000 αυτός ο στόχος. Θα πρέπει να δούμε και κατά πόσο είναι σκόπιμος και κατά πόσον ε, ε, είναι ο κατάλληλος ο μηχανισμός και την αμοιβαιότητα, την αναλογικότητα μάλλον αυτού του μηχανισμού, αν θέλω να χρησιμοποιήσω δικαστική ορολογία. Τώρα, να αναφέρω σε σχέση με όσα ανέφερε ο κύριος αλλά δύο ζητήματα. Για αυτή τη θεώρηση περιοδιαστά πρέπει ο ετών να αποδείξει ε, την πρόθεσή του να παραμείνει στην επικράτεια πολλών ε, πλειώνων κρατών μέλων της Ένωσης. Μα Πώ μπορεί κανείς να αποδείξει την πρόθεση. Να έχουμε ένα πρόγραμμα περιοδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε. Ε, είχε ραντεβού τα οποία, στα οποία παρέστη, είχε νοικιάσει αίθουσε κτλ, Αν έχουμε κάποια πραγματικά στοιχεία, ναι, αλλά ε, πρόθεση, άμα βασιστούμε στι προθέσει, θα μπορούμε να αρνηθούμε να επιτρέψουμε στον οποιονδήποτε να εισέλθει στην ενωσιακή επικράτη. Έχω και μια άλλη ένσταση όμω. για το πώς θα μπορούσε να γίνει κατάχρηση της χρήσης αυτού του μηχανισμού που μας ε, υποβλήθηκε σήμερα. Δημιουργεί λοιπόν θεώρηση που επιτρέπει ουσιαστικά ε, σε μέγιστο διάστημα ενός χρόνου, μπορεί να παραταθεί σε δύο χρόνια, να μπορεί κανείς να μένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέσα σε έξι μήνες πρέπει να μένει το πολύ τρει μήνες σε ένα συγκεκριμένο κράτος μας. Είναι λίγο πολύπλοκο όλο αυτό. Είχαμε δει την πρώτη πρόταση οδηγία του 2001 που ήθελε να δίνει έγκριση έξι διαδοχικών μηνών ε, μέσα σε ένα χρόνο και με μέγιστη παραμονή στο ίδιο κράτο μέλο τριών μηνών. Άρα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα έπρεπε να μένουν τουλάχιστον έξι μήνε εκτό χώρου σέγγιν και μετά να ζητήσουν εκ νέου θεώρηση. Όπω ε, έχει τώρα η πρόταση, δεν προβλέπεται αυτό ο μηχανισμό. Εκτό αν κάνω λάθο βέβαια και δεν ερμηνεύω σωστά αυτό το σύστημα. Άρα, κάποιο ο οποίο πήρε μια θεώρηση, πρώτη θεώρηση για το χώρο σέγγιν δεν χρειάζεται να ξαναβγεί και να ξαναμπεί για να δεύτερη θεώρηση. Άρα αυτό το σύστημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα καθεστώ μόνιμη παραμονής. Κατάλαβα σωστά, κατάλαβα λάθος, μου ξέφυγε κάτι. Διότι αν δούμε και ορεκτικά όπως προβλέπετε αυτό το σύστημα, εγώ καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν ξέρω, ε, μπορεί να κάνω λάθο, βέβαια. Έρχομαι τώρα σε κάποιους ε, τεχνικών παρατηρήσεων για τον κώδικα θεωρήσω για την επεξεργασία των στοιχείων από 15 να πάμε στις 10 ημέρες. Οι αρχές λένε ότι ήδη είναι μικρές προθεσμίες, άρα είναι πτακτική ανάγκη να γίνει αυτό, ερώτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες επισκεπτών που θα πρέπει πλέον να πληρώνουν για την λήψη αυτής της θεώρησης. Μα υπάρχουν πάρα πολλέ κατηγορίε τελικά. Εγώ δεν λέω να είναι δωρεάν η χορήγηση θεώρησης απλά διαρωτώ με αν είναι σκόπιμο να έχουμε αυτό το σύστημα και πάλι το ίδιο τώρα σε ό,τι αφορά τη διάρκεια παραμονής. Θα μπορούσε να ανανεωθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και στο προηγούμενο, για τις θεωρήσεις της περιοδίας δηλαδή. Μέσα σε πέντε χρόνια ξαναξεκινά η διαδικασία από το μηδέν, από την αρχή, χορηγούνται ή δεν θεωρούνται ε, έτους διάρκειας θεωρήσεις πια. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι επιπτώσεις θα έχει, για, ε, με το ε, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το νέο σύστημα. Περιμένω να μου διευκρινίσει τα σχετικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως, επαναλαμβάνω, γίνει πραγματικότητα η μόνιμη παραμονή στο ε, έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά την ιατρική ασφάλιση ταξιδίου, υπάρχουν και εδώ κάποια ζητήματα και ένα τελευταίο ζήτημα, πολύ συγκεκριμένο προς την Κομισιόν πάλι στρεφόμενος. Εδώ είμαι ελαφρώ από τον Λόπεθ Αγγιλάρ. Οργανικά δεν νομίζω ότι είναι αλληλοσυνδεόμενα αυτά τα δύο ζητήματα, περί, ε, θεώρηση περιοδία και κώδικα θεωρήσεων, γιατί η θεώρηση περιοδία είναι μια νέα πρόταση. Για την ανθρωπιστική βίζα, την ανθρωπιστική θεώρηση. Γιατί δεν μα κάνει μια νέα πρόταση Κομισιόν. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την ομάδα Άλτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα έπρεπε να είχα πει ότι είσαστε και σκιώδης εισηγητής της Άλντε. Συνάδελφοι, θα κλείσω τον κατάλογο των εμιλητών. Η τελευταία παρέμβαση ενέπνευσε αρκετούς από εσά να ζητήσετε το λόγο. Θα κλείσω λοιπόν το λόγο τώρα, διότι αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο για τα άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κυρία Ρούσα Τόματιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να ε, συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Ορτεφέ, για την έκθεσή του, στην οποία εστιάζει την προσοχή στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις θεωρήσεις. Ε, η πρόταση ε, παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2014 με στόχο την απλούστευση των ε, διαδικασιών όσων θέλουν ε, να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λίγες μέρες περικόπτοντας το κόστος, διατηρώντας όμως το ίδιο επίπεδο ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεώρηση Σέγγεν ή κάποια άλλη επιστοποίηση που να επιτρέπει παραμονή άνω των 90 ημερών στον χώρο Σέγγεν. Και έτσι οδηγούμαστε σε οικονομική ζημία. Γι' αυτό επικροτώ τη δημιουργία αυτής ε, της ε, νέας ε, θεώρησης που επιτρέπει στους ανθρώπους να βρίσκονται στην περιοχή Σέγγεν πάνω από 180 μέρες χωρίς να θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι. Η καινούρια θεώρηση θα προωθήσει την ε, οικονομική ανάπτυξη και τον ε, τουρισμό καθώς ε, και άλλες δραστηριότητες όπως είναι οι τομείς εστίασης και μεταφοράς. Πρέπει να έχουμε μια καλή θεώρηση, για, ένα καλό σύστημα για τις θεωρήσεις. Θέλουμε να προσελκύσουμε καλλιτέχνες, αθλητές, ερευνητές κλπ. Θέλουμε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο ασφαλείας στα σύνορά μας και μία πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για την Κομισιόν δείχνει το 2012 6,6 πιθανοί ταξιδιώτες από την ε, Κίνα, την ε, Ρωσία, την ε, Ουκρανία χάθηκαν λόγω των επαυτών διαδικασιών για τις θεωρήσεις. Υπάρχει ελπίδα ότι η απλοποίηση θα ενθαρρύνει ε, μεσοαστούς από τι αναδυόμενε οικονομίες να επιλέξουν την Ευρώπη για τις διακοπέ τους αντί για κάποιο άλλο μέρο. Εγώ προέρχομαι από την Κροατία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει σημαντικό αντικτύπο στην οικονομία στο σύνολό της. Ε, θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρισμού ε, επικροτεί την πρόταση, πιστεύει ότι θα βοηθήσει τον τομέα και θα ε, οδηγήσει σε ανάπτυξη ε, στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρώντας και ένα επίπεδο ελέγχου στα λιμάνια, στα αεροδρόμια κλπ. Υπάρχουν όμως κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Για παράδειγμα, θα είναι απαραίτητο το σύστημα να παρέχει επαρκή συντονισμό με τον υπάρχοντα μηχανισμό ασφαλείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα πρέπει να υπάρχει λειτουργικότητα με το σύστημα πληροφόρησης για τις θεωρήσεις και το σύστημα πληροφόρησης Schengen. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ε, παρέκκλησης για κάποια κράτη-μέλη και διμερών συμφωνιών απαλλαγής από τις θεωρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τους συναδέρφους να περιοριστούν σε δύο λεπτά. Παρακαλώ κύριο Σκρουέλ. Θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπρίς Οχτεφέ για το εξαιρετικό έγγραφο εργασίας, το οποίο μας δίνει μια πολύ γερή βάση για ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ο κύριος Οχτεφέ έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι ε, αντιμετωπίσουμε τις εξής περιστάσεις. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι η νομική βάση και το γεγονός ότι υπάρχει τελικά νομικό κενό. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να κάνουμε τους απαραίτητους ε, ελέγχους της κατάλληλες επαληθεύσεις για το αν τελικά οι δικαιούχοι τέτοιων θεωρήσεων όντως τηρούν τις προθεσμίες που προβλέπονται από την νομοθεσία, γιατί αυτή τη στιγμή όντως βρισκόμαστε σε έναν χώρο Σέγγεν χωρίς εσωτερικά σύνορα, άρα χωρίς ε, επαληθεύση συγκεκριμένης παραμονής σε μια χώρα η διέλευση συνόρων. για κάποια άλλα σημεία ενδεχομένω να είχα διαφορετική άποψη. Πάντω ο κύριο Οχτεφέ έχει δίκιο όταν λέει ότι θα πρέπει να δούμε ποιε θα είναι οι συνέπειε από τη νέα αυτή θεώρηση όσον αφορά το ζήτημα τη ασφάλεια. Επίση, έχει δίκιο όταν λέει ότι θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του μηχανισμού αυτού, προκειμένου όντω να δούμε αν θα υπάρχουν θετικέ συνέπειε από οικονομική πλευρά. Και συμφωνώ επίση με τον κύριο Οχτεφέ όταν λέει ότι θα πρέπει η μελέτη αυτή να είναι σαφώς ανεξάρτητη. Ο Ζεχάρ Ντεπρέ έχει δίκιο κι αυτός όταν λέει ότι ενδεχομένως να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι και αισιόδοξοι όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις για την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως όμως να είναι κάπως υπερβολικός όσον αφορά τις επιπτώσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν νομίζω ότι θα αυξηθεί το διοικητικό άχθος με τη νέα αυτή θεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τις συνέπειε για τον τουρισμό, εγώ προέρχομαι από την Πορτογαλία. Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικό τομέα για μα και όντως υπάρχουν έγγραφα τα οποία καταδεικνύουν ότι ε, η θεώρηση αυτή θα μπορούσε όντως να ευνοήσει όχι μόνο τους ε, τουρίστες εκείνους οι οποίοι πρέπει να διέλθουν τα ευρωπαϊκά σύνορα και κάθε φορά που καταφθάουν σε ένα κοινοτικό λιμένα, αλλά θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερη ευνοϊκή θεώρηση αυτή και για τους ίδιους τους ναυτικούς, για το πλήρωμα δηλαδή των ε, διαφόρων πλοίων. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, να δοθεί μια λύση μέσω της ε, θεώρησης αυτής και ενδεχομένω αυτή η θεώρηση περιουδίας να αποτελεί την κατάλληλη απάντηση. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, να πω ότι ε, ελπίζω και εγώ ότι θα μας δώσει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Δεχώστα είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα καταρτισμένος ε, στο ζήτημα αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε και τις δικές του τις εξηγήσεις. Και συμφωνώ κάπως στην σύνεση που δείχνει ο Μπρίς Ορτεφέ, ο οποίος είναι πολύ προσεκτικός με το ζήτημα της ασφάλειας. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση κλειστό οχυρό, αλλά θα πρέπει να καταφέρουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι καλόπιστα επιθυμούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Next is Mrs. Revo Bonifoy. Κύριε Ρεβό Ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο όσον αφορά τις ε, ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Νόμιζα ότι κάναμε κοινή συζήτηση που κάλυπτε και το ζήτημα αυτό. Από ό,τι φαίνεται όμως όχι, επομένως θα ήθελα να πάρω το λόγο αφού μιλήσει ο κύριος ε, Λομπέσα Γουιλάρ. Θα μιλήσω λοιπόν λίγο αργότερα για το ζήτημα της ανθρωπιστικής θεώρησης. Ευχαριστώ. Θέλατε τώρα να μιλήσετε κύριε Λόπη Γουιλάρ. Ναι, λυπούμε που υπήρξε κάποια σύγχυση γιατί τουλάχιστον στο σχέδιο ημερήσια διάταξη προηγείται ο κώδικα θεωρήσεων και μετά η θεώρηση περιοδία, διότι η πρώτη πρωτοβουλία είναι η αναδιατύπωση του κώδικα θεωρήσεων και συμπληρωματικά έρχεται το θέμα της θεώρησης περιοδίας. Άρα τελικά εγώ αυτό το οποίο έκανα ήταν να απαντήσω στα σχόλια και την παρουσίαση του κυρίου Ορτεφέ. Δεν παρουσίασα τα περικόδικα θεωρήσεων. Αν όμω η συζήτηση είναι κοινή, τότε πρέπει να σα παρουσιάσω τα στοιχεία τη δική μου έκθεση. Γιατί έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Για να ε, σας τα μεταφέρω και να μπορείτε κι εσείς να τα ε, ακούσετε και να δείτε ε, αν μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πακέτο. Άρα, να κάνω μια σύνοψη. Δεν είχα καταλάβει, νομίζω ότι θα ήταν το επόμενο σημείο της και αλλά ε, παίρνω κατευθείαν στην παρουσίαση του θέματο. Συνοπτικά λοιπόν, Όπω είπα και πριν, Έχουμε εδώ και κάποιο καιρό ε, συνεργαστεί με τον κύριο Ορτεφέ στο θέμα τη θεωρήση περιοδία ό,τι αφορά την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο και επομένως ε, στο διάστημα αυτό ουσιαστικά ε, βάλαμε σε τροχιά πάλι τα θέματα αυτά και είμαι αισιόδοξο ότι θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε καταρτήσει από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, αυτό που σχεδιάζουμε να κάνουμε είναι να διοργανώσουμε μια ακρόαση εμπειρογνωμόνων ε, τον Ιούνιο στην Επιτροπή μας. Οι εμπλεκόμενοι φορείς λοιπόν θα μας ε, δώσουν ε, τις απόψεις τους. Θα καλέσουμε αυτούς που ενδιαφέρονται περισσότερο για την αναδιατυπωμένη αυτή του κώδικα θεωρήσεων που καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αν θέλουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα της ε, ασφάλειας δικαιοσύνης ελευθερίας. Νομική βάση είναι το άρθρο 77. Άρα, εφόσον υπάρχει σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, Σέγγεν, στο χώρο τη ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο θεωρήσεων και με βάση την προσωπική εμπειρία που είχα μετά από όλες αυτές τις συναντήσεις που είχα μέχρι στιγμής, φαίνεται να είναι ένα άκρος τεχνικό ζήτημα, αλλά δεν είναι. Είναι άκρος πολιτικό και επηρεάζει την καρδιά των σχέσεων μας με τρίτες χώρες. Ουσιαστικά είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει για τα κράτη-μέλη και εφαρμόζεται από τα προξενία των τρίτων χωρών και έχει να κάνει και με την εικόνα που δίνουμε προς τα έξω ως Ένωση. Θέλουμε να προωθήσουμε τις πολιτικές κοινωνικές, ε, επιστημονικές ανταλλαγές και θέλουμε βέβαια και την οικονομική ανάκαμψη να πετύχουμε αυτό το στόχο. Για να μην πω βέβαια ότι υπάρχει και η πτυχή της ασφάλειας. Σημάνθηκε όμως και θέλω και εγώ να το τονίσω. Υπάρχει και ανθρωπιστική πτυχή των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Μιλάμε για ανθρώπους εδώ. Μιλάμε για επικός τρίτων χωρών που χτυπούν την πόρτα, χτυπούν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα συστατικά, όλα αυτά είναι τα κομμάτια του παζλ. Μια, ε, ένας χώρος χωρί χωρίς εσωτερικά σύνορα απαιτεί επιτυχημένο συνορικό έλεγχο ή έλεγχο των εξωτερικών συνόρων που θα ενισχύεται και από μια σωστή πολιτική θεωρήσεων. Έχουμε εδώ τον κώδικα θεωρήσεων που είναι αποτελεσματικός. Από το 2009 ε, χρονολογεί το καθονισμό, ο κανονισμος 10 810-2009 στην απόφαση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και για τις προϋποθέσεις και για τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα προξενία των κρατών μελών της Ένωσης, αντικατέστησε τις λεγόμενες κοινέ προξενικές εγκυκλίους. Άρα οδήγησε σε παγίωση, ενοποίηση και απλούστευση του κεκτημένου. Όμως, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εφαρμογή των διαδικασιών δεν ήταν η βέλτιστη δυνατή. Υπήρξαν ε, ελλείψεις, δυσκολίες, όπως έδειξε η εμπειρία. Θεωρήθηκε λοιπόν σκόπιμο να προταθεί επικαιροποιημένη έκδοση αυτού του κανονισμού προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα που είχαν προκύψει με την αξιολόγηση. Διτά τα προβλήματα. Πρώτον, έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται σωστά από τα προξενία ο κώδικας των θεωρήσεων. Εξωτερική ανάθεση για να είμαι πιο συγκεκριμένος, σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. Ο κώδικας προβλεπόταν ως ένα εργαλείο έσχατης ανάγκης. Αυτό λέει αρχικά ο κώδικας, αλλά στην πράξη έγινε μια κανονική διαδικασία. Και τίθενται ζητήματα που αφορούν και την ποιότητα των διαδικασιών και την προστασία των δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως ε, τις εξουσίες που έχει για να ε, υπάρξει σωστή εφαρμογή του κώδικα. Αυτό σημαίνει ε, κίνηση διαδικασιών επί παραβάση. Αυτό είναι απαραίτητο. Γιατί πρέπει να περιοριστεί αυτή η μαζική εξωτερική ανάθεση που έγινε ουσιαστικά ο κανόνας και όχι εξαίρεση από τα προξενία. Δεύτερον, υπάρχει ένα πρόβλημα κακής ερμηνείας ή παρερμηνείας, ε, πολύ μεγάλη διακριτική ευχαίρεια αν θέλετε ε, στις διαδικασίες. Με αποτέλεσμα να χαθούν κάπου στο δρόμο κάποια στοιχεία ή έλλειψη εκπροσώπησης ε, κάποιων χωρών σε κάποια κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή οι ετούντες θεωρήσεως, οι οποίοι έρχονται ε, και ταξιδεύουν σε άλλα κράτη. Στρέφονται σε κάποιο άλλο ε, κράτος αντί ε, του κράτους που παρόλα αυτά εκπροσωπείται σε εκείνη τη χώρα. Δεν υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των προξενείων. Οι διπλωμάτες δεν συνεργάζονται. Δεν υπάρχει διπλωματική αλληλεπικάλυψη. Και άλλες παρατυπίες εντοπίζονται. Και έχουμε πίσω από όλα αυτά ε, ανθρώπους και τις ιστορίες τους και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε για τις ζωές ανθρώπων. Τα προβλήματα αυτά λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με κοινή προσπάθεια. Και ίσως με την αναδιατύπωση αυτού του κώδικα θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε ε, τη ζωή πολλών ανθρώπων που χτυπούν ε, τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθώντας να εισέλθουν σε αυτήν. Και όχι μόνο με νόμιμα μέσα, αλλά και παράτυπα. Αλλά είναι και πολλοί αυτοί που επαναλαμβάνω ε, νομίμως προσπαθούν και επανειλημμένως για πολύ βάσιμους λόγους να εισέλθουν στην Ένωση για να ε, ασκήσουν κάποια δραστηριότητα. είναι παρατεταμένες, ε, δυσκίνητες ε, και δαπανηρές αυτές οι διαδικασίες και το ε, διαβάζουμε συνεχώς σε όλα τα έγγραφα. Αυτά τα τρία επίθετα έρχονται και ξανάρχονται. Παρατεταμένες, δυσκίνητες, δαπανηρές, συνεχώς αυτά τα τρία επίθετα. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνει τη διαδικασία χωρίς όμως να έχουμε αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια βέβαια. Άρα φυσικά και πρέπει να επικροτήσουμε και να στηρίξουμε την προσέγγιση αυτή. Να έχουμε αυτή την αναδιατυπωμένη εκδοσή του κώδικα που θα επιτυγχάνει μεγαλύτερη ευελιξία Θα έρει τον κανόνα που λέει ότι ο ετών πρέπει να είναι παρόν αυτοπροσώπους να παρουσιάζεται δηλαδή στα προξενικά ε, γραφεία. Να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε δηλαδή τις νέες τεχνολογίες ε, για τον πολύ καλό σκοπό κατάργησης αυτής της ανάγκης, αυτοπρόσωπης παρουσίας ε, σε ένα προξενείο για την θεώρηση. Και τα θα πρέπει να είναι και μικρές προθεσμίες και να έχουμε ένα κοινό κατάλογο των απαιτούμενων εγγράφων. Λήψη τακτιλικών, αποτυπωμάτων περιοχή, κάποια άλλα τεχνικά στοιχεία για τα διάφορε δομογραφίε, ακρονίμια και βέβαια πρέπει να βασιζόμαστε στις, ε, ε, στα αξιόπιστα στοιχεία. Έχουμε και τις λεγόμενες θεωρίες πολλαπλών εσόδων. Αυτή η πρόταση λοιπόν, όπως είπα, πρέπει να υποστηριχθεί για να δούμε Πώ θα προχωρήσουν πω είναι εμπρό. Ολοκληρώνοντα. θα προχωρήσουν προ τα εμπρο Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στι ανθρωπιστικέ θεωρίε που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Με έχει απασχολήσει εδώ και καιρό το ζήτημα αυτό. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι επί ευκαιρία τη αναδιατύπωσης του κώδικα θεωρήσεων θα έπρεπε να δούμε κατά πόσον πρέπει ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι και μπορούμε και πρέπει να κάνουμε κάτι λοιπόν με το εργαλείο αυτό, ώστε να προωθήσουμε τις χορηγήσεις ε, θεωρήσεων ανθρωπιστικών. Και ο λόγος είναι απλός, κατ' Έχουμε 100 θυμάτων ε, στη Μεσόγειο. Θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε ε, την Κομισιόν που δεν κάνει τίποτα, το Συμβούλιο που δεν κάνει τίποτα. Θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε την έλλειψη πολιτικής ε, ή την ε, αναποτελεσματική πολιτική. Υπάρχει δηλαδή και το θέμα αυτό το νομοθετικό. Πιστεύω ότι μπορούμε να και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην χαθούν άλλες ζωές στη θάλασσα. Ναι, ναι, ναι, ολοκληρώνω. Στον σημερινό, στον ισχύοντα κώδικα θεωρήσεων υπάρχουν διατάξει που επιτρέπουν την έκδοση τροπιστικών θεωρήσεων, δεν είναι σαφή οι λόγοι όμω και οι προποθέσει. Υπάρχει το ενδεχόμενο, η δυνατότητα παρέκκληση ε, των κανόνων επιλεξιμότητα όταν μιλάμε για ανθρωπιστικέ ανάγκε. Δεν υπάρχει όμω διασύνδεση με τον κανόνα ότι αυτό αποτελεί λόγο ε, βάσιμο για την έκδοση και τη χορήγηση ανθρωπιστικής θεώρησης. Υπάρχουν όμως ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και το άρθρο βέβαια 19 και 25 του κώδικα που λέει ότι θα μπορούσε να εκδοθεί θεώρηση περιορισμένη ανταφική ισχύω αν θεωρείται για ανθρωπιστικού λόγου αυτό απαραίτητο από ένα κράτο μέλο. Μα αυτό ε, το κάνει η Βραζιλία για τη Συρία. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Να εκδώσουμε λοιπόν σε έκτακτες τέτοιες περιστάσεις σε ανθρωπιστικές θεωρίες. Ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Συνεργασία μεταξύ προξενείων. Διευκόλυνση της διαδικασίας. Να είναι πιο βραχίες ε, οι διαδικασίες και λιγότερο δυσκίνητες και παρταμένες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τον κώδικα θεωρήσεων. Φυσικά και θα συνεργαστώ με τα προθυμία και με τον κύριο Ορτεφέ και με τους υπόλοιπους όδε και όλους του τους όλων των πολιτικών ομάδων. Μέσω των προβληματισμών των απόψεών τους πιστεύω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη και από τους δύο εισηγητές που άλλαξα τη σειρά ε, στην αρχή. Εγώ φταίω. Ζητώ συγγνώμη. Θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Ορτεφέ να απαντήσει στη σύνοψη του κυρίου Λοπές Αρκιλάρ. Και κατόπιν να περάσουμε στο θέμα των θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Σας παρακαλώ να περιοριστείτε όλοι οι ομιλητές σε ένα με δύο λεπτά, διότι πρέπει να ακούσουμε απαντήσεις της Κομισιόν σε πολλά θέματα ουσίας που ακούστηκαν. Και μετά, μην ανησυχείτε, δεν έχω ξεχάσει τους ε, τρεις τελευταίους ομιλητές. Θα μπορούν έτσι να απαντήσουν ε, στο κυρίως σώμα της συζήτησης και στο τέλος θα ακούσουμε την Κομισιόν που θα απαντήσει σε όλους. Ο κύριος Ορτεφέ πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Μπέκερ δεν μπορεί να παραστήσει συνεδρίαση, θα έπαιρνε κανονικά το λόγο. Ο εισηγητή, θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποιε από τι ανησυχίε που ακούσαμε. Ο κύριο Μπέκερ προφανώ θέλει να ευχαριστήσει τον συνάδελφο Λόπε Αγκουιλάρ και τους συνεργάτες του για την πολύ καλή συνεργασία που είχαν εγκρίνει την προσέγγιση του εισηγητή και συμφωνεί και αυτός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξίας στις προξενικές αρχές όσον αφορά τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν ως δικαιολογητικά και όσον αφορά το ζήτημα της αυτοπρόσωπης παρουσίας των ετούντων. Μέσω των προξενικών αρχών θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε φορά που εκπροσωπούνται χώρες σε τρίτες χώρες και να μειωθούν επίσης και οι προθεσμίες που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις που χορηγούνται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστεί κ. Μπέικερ τον Χουάν Φερνάντο, διότι και αυτός θεωρεί ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή να υπονομεύσει την γενικότερη κλασική διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων. Επίσης, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα άτομα τα οποία θα πάρουν μια τέτοια θεώρηση, ότι θα παραμείνουν στο κράτο μέλος το οποίο έδωσε αυτή τη θεώρηση. Για παράδειγμα, δεν θα είμαστε σε θέση να δούμε τελικά αν τα άτομα αυτά θα παραμείνουν στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο κάνουν αίτηση. Πώς μπορεί δηλαδή ένας υπάλληλος ασφαλείας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει τις επαληθεύσεις που πολλές φορές γίνονται σε διάστημα 15 ημερών από τους υπαλλήλους των προξενικών αρχών. Πρέπει να αποχωρήσω κύριε Πρόεδρε, έχουμε στη Γαλλία εκλογές σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο σε 15 περίπου ημέρες, επομένως πρέπει να επιστρέψω στη Γαλλία. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε, και το τονίζω αυτό, μία μελέτη αντικτύπου. Καταλαβαίνω ότι έχει κάποιες επιφυλάξεις προς αυτό ο κύριος Λόπες Αγκουιλάρα αλλά προβλέπεται άλλωστε μια κρόαση όπως είπαμε τους επόμενους μήνες. Θεωρώ ότι όντως πρέπει να έχουμε τέτοια κρόαση και θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση περισσότερο στην εμπειρογνωμοσύνη όσων προτείνουν τη νέα αυτή νομοθεσία και όσων πρόκειται να αποφεληθούν από τη νέα αυτή νομοθεσία. Σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν που πρέπει να αποχωρήσω γρήγορα και προφανώς εφόσον έχετε ερωτήσεις μπορείτε να τις απευθύνετε στο γραφείο μου και θα φροντίσω να απαντήσω το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ και πάλι συγγνώμη που άλλαξα τη σειρά των θεμάτων. President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση του κώδικα θεωρήσεων θα μας επιτρέψει να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ελκυστική, διατηρώντας την εκαιρότητα του χώρου Σέγγεν. Προφανώς δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι απόρθητο φρούριο, αντίθετα θέλουμε μια ανοιχτή Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα πιο συγκεκριμένα για τις θεωρίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Λόπες Αγγουλάρη για τα όσα είπε πριν από λίγο. Συμφωνώ με τα συμπεράσματα της μελέτης η οποία θα μας παρουσιαστεί σε λίγο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό ανθρωπιστικών θεωρήσεων, άλλωστε αυτό προβλέπεται και από τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους πρόσφυγες ή τους ετούντες άσυλο. Ένα 90% των ανθρώπων που ζητούν διεθνή προστασία συνήθω διακινδυνεύουν την ίδια τη ζωή του προκειμένου να έρθουν στην Ήπειρό μα. Και σήμερα το πρωί ακόμα είδαμε απέσιε εικόνε στι ειδήσει, στι τηλεοράσει μα από ανθρώπου που χάσαν τη ζωή του προσπαθώντα να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να θελοτυφλούμε όσον αφορά την, τον πραγματικό λόγο του προβλήματο. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσημοι διάβλοι για του ανθρώπου αυτού προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να έχουν νόμιμη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει αυτό να γίνει υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του νέου κώδικα θεωρήσεων να προβλέπονται αυτοί οι νέοι επίσημοι μηχανισμοί. Δύο ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένω να μα απαντήσει, ενδεχομένω και όχι. Πρώτη ερώτηση, απευθυνόμενη κυρίω στο Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα κινούνται στα πλαίσια των κρατών μελών. Θα έχουμε δηλαδή μια συμφωνία. Και δεύτερη ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα υποχρεωτικό στα πλαίσια του κώδικα θεωρήσεων όσον αφορά τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις και ο ίδιος ο Επίτροπος Αβραμόπουλος είχε δεσμευτεί ως προς αυτό. Ο κύριος Κουέλιο θα απαντήσει. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Αγγιλάρ ότι τον ευχαριστώ για τη δουλειά που έχει κάνει και συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις του σχετικά με το outsourcing, την εξωτερική ανάθεση. Νομίζω ότι είναι τροπή ότι κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα με κακό τρόπο. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ο κώδικας θεωρήσεων να είναι συνεπής, να είναι ο ίδιος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη για τον εθνικό πυλώνα των θεωρήσεων. Θα πρέπει να είναι συνεπής ο κώδικας και να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο, όπως είπε και ο Φερνάντο. Ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητο να έχουμε τους μηχανισμούς για να ελέγχουμε την εφαρμογή του. Όπως είπε ο κύριος ε, Αγκυράρ, θα πρέπει να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τους κανόνες αυτούς. Ο, ο νέος μηχανισμός αξιολόγησης Schengen θα επιτρέψει τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο από ποτέ και πιστεύω ότι μετά από τον πρώτο γύρο θα μπορέσουμε να εξετάσουμε εάν απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία. Θα ήθελα επίσης ε, να ε, τονίσω τη σημασία της πρότασης για το VIS, ε, το σύστημα πληροφόρησης για τις θεωρήσεις. Δεν είναι συχνά ε, που βλέπουμε προτάσεις για την χρήση συστημάτων που ήδη έχουμε. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ε, τα εργαλεία αυτά, πιστεύω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο το VIS. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κάρλος. Και τώρα για το σύνολο της συζήτησης. Πρώτα Σκά Κέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους εισηγητές μας ε, για το θέμα αυτό. Σημεριζόμαστε την άποψη που έχει εκφραστεί και νωρίτερα ότι θα πρέπει να είναι πιο εύκολο για τους ταξιδιώτες να έρχονται στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να ε, προσθέσω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τους ε, πλούσιους ανθρώπους. Και οι φοιτητές χρειάζονται ένα απλουστευμένο σύστημα έκδοσης θεωρήσεων. Συμμεριζόμαστε πολλές από τις θέσεις της, ε, των προτάσεων της Κομισιόν. Δεν θέλω να αναφερθώ στα επιμέρους σημεία. Συμμερίζομαι όμως ε, και την ανησυχία του εισηγητή για την εξωτερική ανάθεση και ε, δεν αρκεί απλά να διαγραφεί η διάταξη. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί όσον αφορά το θέμα αυτό. Και το πιο σημαντικό κομμάτι για μας είναι η θεώρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν, πολύ λίγα κράτη-μέλη την χρησιμοποιούν. Μπορούμε όμως να τη χρησιμοποιήσουμε για να επιτρέπουμε στους ανθρώπους ε, να έχουν νόμιμη και ασφαλή ε, είσοδο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, χρειάζεται να ε, έχουμε ένα σωρό μελέτες. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Αγγιλάρο ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε την προσέγγιση στο θέμα αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα που μπορούμε να εξετάσουμε. Η Βραζιλία την χρησιμοποιεί με πολύ αποτελεσματικό τρόπο για τους Σύριους πρόσφυγες. Είναι σαφές ότι όταν κάποιος ε, φεύγει από τη Συρία έχει πολύ καλούς λόγους για κάτι τέτοιο. Ίσως ε, λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε την ε, πιθανή πρόσβαση τέτοιων ανθρώπων χωρίς θεώρηση καθόλου. Επίσης θα απαιτηθεί η θεώρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βενπέργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ στον χρόνο ομιλία. Πάντα στην ώρα μου Έχουμε και τηρώ το χρόνο ομιλία. Ήθελα να αναφερθώ στην θεώρηση ανθρωποστικού χαρακτήρα, αλλά ευχαριστώ, θα μιλήσω ε, και για το θέμα που συζητάμε τώρα ή θα μου δώσετε χρόνο ομιλίας για το σημείο 6 ε, ή να τα πω τώρα. Φαίνεται ότι υπάρχει παρανόηση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε. όσον αφορά τον κώδικα θεωρήσεων, νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει τελείως την πτυχή της ασφαλείας. Αυτό είναι το μεγάλο μου ερώτημα. Έχουμε εξετάσει το θέμα αυτό. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την ασφάλεια. Διαφωνώ με την διαγραφή της απέτησης για ιατρική ασφάλιση. Γιατί? Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις κινδύνου για όλους τους ετούντες για να ανακαλύψουμε και τους παράνομους και βλέπουμε ότι εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί άνθρωποι τους οποίους δεν ελέγχουμε, βλέπουμε και τρομοκράτες. Επίσης, ε, πολλοί άνθρωποι μένουν παραπάνω από όσο τους επιτρέπει η θεώρηση. Πάντως, η βασική μου ανησυχία είναι το θέμα της ασφαλείας και ελπίζω να μου δώσετε και το λόγο στο σημείο 6. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Μιέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις ε, σχετικά με την θεώρηση περιοδίας. Νομίζω ότι οι ίδιοι επιχειρηματίες και άλλοι άνθρωποι έχουν πολλούς τρόπους ε, να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι με ένα τέτοιο νέο σύστημα μόνο περισσότερους κινδύνους θα έχουμε. Η ε, θεώρηση περιοδίας ε, θα είναι πολύ εύκολο να παραβιαστεί και έτσι θα έχουμε ανθρώπους που θα κινούνται στον ε, χώρο Σέγγεν ε, χωρίς έλεγχο και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε διπλασιασμό των λαθρομεταναστών ε, στα εδάφη μας και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε. Υπάρχει λοιπόν εδώ σημαντικός κίνδυνος όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Και ποιος λέει ότι μόνο τουρίστες και συνταξιούχοι θα χρησιμοποιούν αυτή την βίζα και όχι το Ισλαμικό κράτος. πόσο μάλλον εάν παραμείνουν παραπάνω από όσο τους επιτρέπει η θεώρηση και αρχίσουν να τριγυρνάνε στα διάφορα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποτρέψουμε τέτοιες καταχρήσεις και να προστατεύσουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλους δύο μιλητές έχουμε. και η προσκεκλημένη μας θα μου επιτρέψει να τους ακούσουμε πρώτα. Κυρία Στίβενς, είναι σκιώδης εισηγήτρια, γι' αυτό ήθελα να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, το ECR επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιέχει κάποια πολύ καλά στοιχεία που ε, κάνουν ε, λιγότερο χρονοβόρα την εφαρμογή του συστήματος για τις θεωρήσεις. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής ε, αίτησης και χρήσης ε, σύγχρονων ε, συστημάτων επικοινωνίας όπως είναι το Skype για συνεντεύξεις. Έτσι θα διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες και θα διευκολυνθούν οι οικογενειακές επισκέψεις και ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από κάποιες ε, μικρές προσαρμογές έχουμε εντοπίσει τέσσερα θέματα στην παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και στο έγγραφο εργασίας ε, του εισηγητή. Η κατάργηση της απέτηση για ιατρική ασφάλιση. Η κατάργηση για την απέτηση υποβολής εγγράφων ε, για τους ε, συχνούς ταξιδιώτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο VIS. Οι νέες ε, λεγόμενες χρυσές βίζες στα εξωτερικά σύνορα και τέλος την πρόθεση του εισηγητή να κινηθεί προς τη δυνατότητα έκδοσης θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Και τα τέσσερα αυτά σημεία που μόλις ανέφερα ανησυχούν το ECR, ωστόσο λόγω περιορισμένου χρόνου θα επικεντρωθώ στα δύο τελευταία σημεία. Πρόεδρε, συνάδελφοι, καταρχάς όσον αφορά τις λεγόμενες χρυσές θεωρήσεις. Ζητήθηκε από την Τουρκία να ευθυγραμμίσει την πολιτική θεωρήσεών της με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταργήσει την έκδοση θεωρήσεων στα σύνορα, πράγμα που έκανε. Γι' αυτό φαίνεται περίεργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να θέλει να επανεισάγει το σύστημα αυτό, για παράδειγμα στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στο πιλωτικό πρόγραμμα. Έτσι ένα κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα αυτόνομα και χωρίς προϋποθέσεις να αποφασίζει σχετικά με μια τυχαία ομάδα ανθρώπων για τους οποίους θα εκδίδει θεωρήσεις για το σύνολο του χώρου Σέγγεν. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους εάν δεν έχουμε τις σωστές διαδικασίες επαλήθευσης και εάν δεν έχουμε την απαραίτητη τεκμηρίωση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, ολόκληρα τμήματα του κώδικα θεωρήσεων ε, σχετικά με την επαλήθευση της πρόθεσης των ταξιδιωτών να εγκαταλείψουν πάλι τον χώρο Σέγγεν. Επίσης, ε, με ανησυχεί κάπως η θέση του εισηγητή ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την δυνατότητα χορήγησης θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω πολύ καλά ότι αργότερα θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μετά την παρουσίαση της μελέτης, ωστόσο, θα ήθελα ήδη τώρα να δράξω την ευκαιρία να σας πω ότι πιστεύουμε ότι ο κώδικας θεωρήσεων δεν είναι το απαραίτητο εργαλείο για την επανεκατάσταση των προσφύγων. Ευχαρίστω να συζητήσω το θέμα αυτό, αλλά ε, όχι ταυτόχρονα με την συζήτηση για την ε, μεταρρύθμιση του ενωσιακού κώδικα θεωρήσεων. Ε, και επίσης μας αποσχολεί το θέμα της θεώρησης περιοδίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, γενικά θέλω να ακούμε τους κοιόδες εισηγητές στην αρχή μιας συζήτησης. Όταν όμως ε, δεν βρίσκονται εδώ στην αρχή της ε, συζήτησης, αν γνωρίζετε ότι θα έρθετε, σας παρακαλώ να μας ενημερώνετε για να το γνωρίζουμε. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Σκοράου, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Καταρχάς, να συγχαρώ τον εισηγητή Λόπε Αγκουιλάρα για την εργασία την οποία έκανε και συμφωνώ με πάρα πολλές από τις παρατηρήσεις του. Κατά την άποψή μας, οποιαδήποτε απλούστευση θα πρέπει να επιδοκιμαστεί, όσον αφορά δηλαδή τον νοσιακό κώδικα θεωρήσεων, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε καλύτερη εφαρμογή του και καλύτερη ε, αποτελεσματικότητα μέσω του κώδικα αυτού στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχουν ε, μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς σε καθημερινή βάση βλέπουμε πάρα πολλές τραγωδίες στην Μεσόγειο πολλές παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάπως αντιφατικές. Μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος επιμερισμός του άκθους αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά την διεκπαιρέωση των θεωρήσεων. Από την άλλη όμως ενδεχομένως οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις να αποτελέσουν μια παράκαμψη του ίδιου του κανονισμού του Δουβλίνου και ήδη στα πλαίσια του κανονισμού του Δουβλίνου νομίζω ότι δεν έχουμε τον καλύτερο δυνατό επιμερισμό των αρμοδιοτήτων όσον αφορά την, τον νοσιακό κώδικα θεωρήσεων. Επίσης, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε όντως ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις θεωρήσεις αυτές ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι θα, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να αυξηθεί εξαιτίας των θεωρήσεων αυτών των ανθρωπιστικών ο αριθμός των μεταναστών αυτών που θα θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μέσο αυτό. Σίγουρα θα πρέπει να βασιστούμε σε ένα σύστημα αλληλεγγύης, σε ένα σύστημα ευθύνης, όλα όμως θα πρέπει να διέπονται και να κανονίζονται στα πλαίσια του νοσιακού κώδικα θεωρήσεων. Όσον αφορά τώρα τη θεώρηση περιοδίας, νομίζω ότι το μέσο αυτό είναι θετικό. Όντως θα δώσει τη δυνατότητα σε ορισμένε κατηγορίε πολιτών από τρίτε χώρε να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπο πιο εύκολα. Αναφέρομαι αυτή τη στιγμή σε καλλιτέχνε, σε φοιτητέ, σε ερευνητέ, σε σπουδαστέ, ακόμα και σε επιχειρηματίε. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μέσο αυτό. Νομίζω ότι θα δημιουργήσει ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλεια. Αλλά πρέπει εμεί να το προασπίσουμε αυτό, πρέπει εμεί να το διασφαλίσουμε αυτό, όπω είπε ο κύριο Οχτεφέ. Δεν θα πρέπει επίσης να γίνει κατάχρηση του συστήματος αυτού. Τώρα, το κατά πόσο θα καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί να συμβάλλουν οικονομικά στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι όντω θα το κάνουν αυτό και δεν νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλούς τρομοκράτε οι οποίοι θα παρουσιαστούν ως καλλιτέχνε και θα προσπαθήσουν κατά αυτόν τον τρόπο να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να είμαι ειλικρινής, είμαι κάπως απελπισμένος. Δεν είναι, τα, είναι το φόρτε μου τα μαθηματικά, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον 25 σημαντικά θέματα και ερωτήματα ετέθησαν και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ή πόσο χρόνο μου δίνεται τέλος πάντων για να απαντήσω. Πρόεδρος, θα γίνει και μια συζήτηση στη συνέχεια το να είναι επελπισμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια ενδιαφέρουσα είδη. Άλλωστε και στην περιγραφή της εργασίας μας είναι μέσα ότι πρέπει να σας απελπίζουμε. Αλλά απαντήστε έστω στα βασικά ερωτήματα που έθεσαν οι εισηγητές. Αν μπορείτε. Δείξτε δημιουργικότητα και φαντασία. 8 με 9 λεπτά μπορώ να σας δώσω. Είμαι βέβαιος ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσετε. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε μία ακόμη περαιτέρω ανταλλαγή απόψε για αυτό το θέμα. 16 και 17 Ιουνίου θα έχουμε και ακρόαση. Η κατάθεση τροπολογιών 17 Ιουλίου, κατάθεση τροπολογιών 3 Σεπτεμβρίου και 13 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή, άρα θα επακολουθήσουν και άλλοι γύροι συζήτησης. Λυπούμε που δεν σας περιορίζω στο χρόνο, αλλά έχουμε και μία προσκεκλημένη. Θα σας δώσω 8-9 λεπτά. 8-9, αν δεν μπορείτε να κάνω και 10 θα δούμε. Αν θέλουν να σας ρουφήξουν το αίμα, <laughs> θα σας δώσω και παραπάνω χρόνο. Προσπαθήστε όμως να είστε πιο ε, περιεκτικός, γιατί σίγουρα ήταν πολλά τα ερωτήματα και τα έχω καταγράψει και εγώ, οπότε θα τσεκάρω. Πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, είστε πάρα πολύ ευγενικό. Δεν ξέρω αν μειώθηκε η απελπισία που ένιωθα πριν, αλλά τέλος πάντων. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω του συζητητέ και του σκιώδει με τι πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει που είχαμε επί των δύο αυτών προτάσεων. Νομίζω ότι και οι δύο εκθέσει ή έγγραφα εργασία αποτελούν καλή βάση για το περαιτέρω έργο που έχουμε να επιτελέσουμε πάνω στην πρόταση της Κομισιόν. Καταρχάς θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον κώδικα θεωρήσεων. Με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ συμφωνεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη βασική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, όπως αυτό της εξωτερικής ανάθεσης, για το οποίο ακούσαν παρεμβάσεις βουλευτών που λένε ότι είναι πάρα πολύ ε, κακό και τεράστιο πρόβλημα η εξωτερική ανάθεση. Δεν το πιστεύουμε εμείς αυτό. Θεωρούμε ότι η εξωτερική ανάθεση είχε πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο ιδίω σε ό,τι αφορά τους ετούντες. Γιατί είναι πιο κοντά πλέον ε, στον ετούντα αυτά τα γραφεία δεν αρκεί το προξενείο στην πρωτεύουσα μια τρίτη χώρα στι μεγαλύτερε χώρε ή στι ε, πρωτεύουσε. Άρα, ε, μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται αφεαυτού πρόβλημα εξωτερική ανάθεση. Στην αναδιατυπωμένη έκδοση όμως πρότασή μα μας την υποχρέωση των κρατών μελών να αναφέρουν ετησίω τι γίνεται με τη χρήση και την παρακολούθηση της εξωτερική ανάθεσης των, ε, των ε, εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. Αυτή η υποχρέωση δεν εμπεριέχεται στον ισχύοντα κώδικα. Με το νέο μηχανισμό αξιολόγησης θα μπορούμε λοιπόν να διαπιστώσουμε καλύτερα αν λειτουργεί σωστά και συνάδει με τις νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις η εξωτερική ανάθεση. μπορούσα τώρα να μιλήσω λίγο για τις θεωρήσεις περιοδίας και καταλήγοντα, θα μιλήσω εν συντομία για τι θεωρήσει ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ο συγκεκριτή του εγγράφου εργασία εγείρει πράγματι πολύ δικαιολογημένα ερωτήματα και ζητήματα. Για να είμαι πολύ σύντομο, θα μπορούσα να πω εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε πολύ καλέ απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Ο εισηγητή έθεσε το ζήτημα του κατά πόσον δημιουργούμε ε, ένα εργοστάσιο ε, φυσικού αερίου, Ιουζίν Αγκάζ. Υπάρχουν πολλοί πολίτες που έχουν νόμιμο θεμητό ε, συμφέρον να έρθουν στην ε, επικράτεια του Σέγγεν και να παραμείνουν για παραπάνω από 90 ημέρες. Μπορεί να είναι επιστήμος, μπορεί να είναι καλλιτέχνης. Δεν το αφισβητούμε λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον ή συμφέρον. Δεν έχουμε όμως σήμερα ένα νομικό πλαίσιο που να τους το εξασφαλίζει αυτό. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δουλεύουν για το Σεκ Σολέ, για παράδειγμα. Για αυτούς εκδίδεται μια ειδική βίζα από 9 μήνες έως ε, ένα χρόνο. Τέσσερις θεωρήσεις ουσιαστικά. Αλλά αυτό δεν εφηγραμμίζεται με το και εκτιμένο. Σαν εφόσον χρειάζονται τέσσερις αιτήσει και τέσσερις φορές να ελεγχθούν αυτές οι αιτήσει από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Θέλουμε αυτό να το αντικαταστήσουμε με μία εννέα θεώρηση που θα καλύπτει ένα έτος το πολύ. Και από πλευρά νομική βάση, κύριε Πρόεδρε, βέβαια, θα μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά στη συνθήκη τη Λισαβόνα, ο περιορισμό τη βραχία παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τρει μήνες έχει διαγραφεί, έχει απαλληφθεί. Και αυτό ακριβώς για να ρυθμιστούν ε, τα στήματα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν στο χώρο Σέγγεν και να κυκλοφορούν εντό Ένωσης για μεγαλύτερο διάστημα πέραν των παραδοσιακών τριών μηνών. Άρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμφίβολα, υπάρχει νομική βάση Έπειτα ετέθη το ζήτημα της μελέτης αντικτύπου. Ζητήθηκε μια νέα μελέτη αντικτύπου. Θα πρέπει να έρθω σε δημερή επαφή με τον εισηγητή για να του εξηγήσω ότι αναφέρεται στην τρέχουσα μελέτη αντικτύπου που ε, έχει να κάνει με τις αυτές προτάσεις. Φυσικά και μια μελέτη αντικτύπου πρέπει να βασίζεται κατά το δυνατόν σε αποδεικτικά στοιχεία εμείς απευθυνθήκαμε σε εκπροσώπους των διαφόρων κλάδων και του ζητήσαμε να μας πούν ποιο θα ήταν το κόστος από τη μη ύπαρξη θεώρησης περιοδίας. Χρησιμοποίησαμε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία στη μελέτη. Δεν είναι όμως ε, τα μόνα, γιατί δεν μας τα επαγορεύουν ε, οι εμπλεκόμενοι, αυτά που θα γράψουμε στη μελέτη αντικτύπου. Έχουμε λοιπόν και πολλά άλλα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποίησαμε σε αυτή τη μελέτη αντικτύπου και με πολύ μεγάλη μου χαρά θα σας τα εξηγήσω κύριε Ορτεφέ, μάλλον στον κύριο Ορτεφέ που δεν είναι πλέον παρόν, θα τα εξηγήσω διμερώς. Άρα δεν νομίζουμε ότι απαιτείται νέα μελέτη αντικτύπου. Η πτυχή της ασφάλειας τώρα. Είπαν ότι ανοίγει παράθυρο ή πόρτα στις ελαφρομετανάστες ε, η θεώρηση περιοδίας. Θα πρέπει να δούμε τους όρους όμως που πρέπει κανείς να ε, πληρεί για να πάρει αυτή τη θεώρηση περιοδίας. Είναι πολύ πιο αυστηρή η όρη πολύ πιο δύσκολο μπορεί κανείς να το εκπληρώσει σε σχέση για παράδειγμα με την απόκτηση μιας κανονικής θεώρησης Σέγγεν. Αν κάποιος θέλει να εξαπατήσει και να μπει ε, με τη βίζα αυτή και μετά είτε να εξαφανιστεί είτε να μείνει για περισσότερο χρόνο, θα το προσπαθήσει με την κανονική βίζα Σέγγεν και δεν θα επιλέξει τη διαδικασία της αποκτήσης μιας θεώρησης περιοδίας. Και να πω εν παρόδο ότι πάντα στο θέμα της ασφάλειας Σήμερα, επειδή υπάρχουν διμερείς συμφωνίες, τα είπε και ο κ. Σαρτεφέ, μπορούν κάποιοι να παραμείνουν α, σε, ε, για όσο χρονικό διάστημα θέλουν. Υπάρχουν συμφωνίες που ε, υπεγράφησαν το 1950-1960. Μπορεί να μπορούν να μένουν και για 63 μήνες για παράδειγμα, με βάση ε, μία βίζα βραχίας παραμονής. Είναι ένα σύστημα που πλέον δεν έχει καμία λογική, αφού έχουμε την κοινή πολιτική θεωρήσεων. Έχουμε προαιώνιες συμφωνίες διμερείς, δεν μπορούν αυτές να χρησιμοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν λέμε βέβαια, ούτε καταγγέλουμε αυτές τις μέρες μέσα, απλά να διαγραφεί λέμε η διάταξη που λέει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να επιμηκύνει την παραμονή στο χώρο Σέγγεν για μια περίοδο που ορίζεται στη διμερή συμφωνία με βάση τις παλαιές διμερή συμφωνίες που έχουν όπως είπα συναυθεί πριν καν αρχίσει να λειτουργεί ο χώρος Σέγγεν. Άρα σε σχέση και με το πρόβλημα των εξωτερικών σχέσεων πρέπει να πω ότι περισσότερες τρίτες χώρες δεν συμβουλεύουν τους ταξιδιώτες υπηκός των χώρων να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Οι Άπωνες, οι Αμερικανοί. Τους λένε άμα θέλετε να πάτε σε μια χώρα του χώρου Σέγγεν για τρεις μήνες να πάτε. Ενώ οι διμερείς προβλέπουν μεγαλύτερο διάστημα. Άρα, εάν δεν καταγγείλουμε λοιπόν τις συμφωνίες και απλά περιορίσουμε αυτή ε, τη διάταξη στο 20 παράγραφος 2, δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάποιο, κάποια τραγωδία με τις τρίτες χώρες εν γέννη. Μια τελευταία λέξη τώρα για τις θεωρίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξτάζει το ενδεχόμενο της εξέβρισης κάποιων νομικών οδών που άτομα που χρήζουν προστασία θα μπορούσαν να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την επανεγκατάσταση Να μην μιλάμε όμω για βίζε ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ε, ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αλλά για άδειε παραμονή ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Πέρμιτ και όχι βίζα. Γιατί θα μπορούσε κανεί να πει ότι με την θεώρηση Σέγγεν καλύπτεται το πρόβλημα. Όχι. Δεν συμφωνούμε. Οι θεωρήσει Σέγγεν αφορούν βραχίε παραμονέ. αν κάποιο χρήζει προστασία δεν εντάσσεται σε, αυτή την, σε αυτό το κόνσεπτ γιατί ε, χρήση προστασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και όλο ο τρόπο που λειτουργεί η θεώρηση έγκαιν δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση. Αν κάποιο θέλει να έρθει για, μια, ε, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, υποβάλλει την αίτησή του στο κράτο μέλο, του αν ο βασικό του προορισμό. Όμω, αν κάποιο χρειάζεται προστασία, αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να επιλέξει το κράτο μέλο που μπορεί να του παράσχει τα υψηλότερα επίπεδα προστασία και να πει όμω εκεί κάνω την αίτηση και τον, πρέπει να τον δεχτούν. θα πρέπει να ορίσουμε μετά ποσοστώσεις ε, για θεωρήσεις έγκαιν ή μπορούν όλοι, όλος ο κόσμος να υποβάλει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος θεώρηση έγκαιν και ε, αίτηση για, για θεώρηση και να την πάρει. Εμείς δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης του κώδικα θεωρήσεων μπορεί να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν κάποιος, κάπως πιο σοβαρό το ύφος της παρέμβασής σας από ότι στην συζήτηση πριν. Νομίζω ότι αντοκατοπτρίζεται την σοβαρότητα του θέματος. Θα ήθελα να προγραμματίσουμε άλλη μία ανταλλαγή απόψεων. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να επιστρέψετε όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Θα έχουμε τώρα συζήτηση για τις θεωρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Πάντως με τις απαντήσεις σας δώσατε νομίζω ενάψματα για ε, επιπλέον ερωτήσεις. Θα προγραμματίσουμε λοιπόν άλλη μία συζήτηση για τον κώδικα θεωρήσεων. Θα συζητήσουμε βέβαια τώρα το θέμα αυτό, αλλά όχι στο πλαίσιο της Επιτροπής. Θα προγραμματίσουμε λοιπόν μια σχετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που προσπαθήσατε να απαντήσετε σε όσο γίνεται περισσότερες από τις ερωτήσεις αυτές. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορέσατε να απαντήσετε σε όλες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους συζητητές και τους σκιώδεις συζητητές. Συνάδελφοι, τώρα προχωράμε στο σημείο 6. Θεωρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, επιλογή ή υποχρέωση. Την παρουσίαση θα κάνει η κυρία Ούλα Ιπεν Γένσεν, που είναι ανεξάρτητη νομική ερευνήτρια σύμβουλος με έδρα τη Δανία. Η μελέτη που θα μας παρουσιάσει σήμερα τη συζητήθηκε από την ΛΥΜΠΕ και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών. Κυρία Υπενγέννης, να έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να σας παρουσιάσω την μελέτη για τις θεωρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Είναι τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Αυτή τη μελέτη είναι να σα παρουσιάσουμε τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης και να επικεντρωθούμε σε κάποιε από τις τροποποίησεις που μπορούν να γίνουν στον κώδικα θεωρήσεων. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις θεωρήσεις έννοια ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον κώδικα θεωρήσεων, η θεώρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα, έχει περιορισμένη εδαφική ισχύ, δεν ισχύει δηλαδή για όλα τα κράτη-μέλη. Και η νομική βάση είναι το άρθρο 25.1, όπου ε, καλύπτονται οι παρεκκλήσεις από τις απαιτήσει για τις ε, θεωρήσεις Schengen. Και στο άρθρο 19.4 έχουμε επίσης παρεκκλήσεις ε, σχετικά με τις προϋποθέσεις Σύμφωνα με το 25.1 λοιπόν έχουμε διάφορες θεωρήσεις ε, που πρέπει να εξετάζονται. Οι θεωρήσεις περιορισμένης ε, ταφικής ισχύους λέγονται και θεωρήσεις LTV. Καταλαβαίνω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Σας κοιτάξουμε γρήγορα τον ορισμό της θεώρησης ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην μελέτη και κατά διάρκεια της ε, παρουσίασής μου για να καλύψουμε την ε, έκδοση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους ε, και λόγω κάποιων διεθνών συνθήκων. Και ας περάσουμε τώρα στα βασικά συμπεράσματα της μελέτης. Πρώτα να σας κάνω μια επισκόπηση των δύο βασικών συμπερασμάτων. Το πρώτο είναι ότι ο κώδικας θεωρήσεων είναι ασαφής και δεν προβλέπει ξεχωριστή διαδικασία για τις θεωρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, κάτι που ήδη επεσήμαναν κάποια μέλη του Κοινοβουλίου. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει διάφορα σχετικά καθεστώτα ανθρωπιστικών θεωρήσεων, αλλά διστάζουν να στηρίξουν μια ευρωπαϊκή λύση. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο συμπέρασμα, στην σελίδα 24 της μελέτης θα βρείτε τον σχετικό πίνακα. Το διάγραμμα αυτό ε, δείχνει μία ασαφή διαδικασία και πολύπλοκη. Αυτή λοιπόν η παρούσα διαδικασία για τις θεωρήσεις αυτές όπου εξετάζονται θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα σε μια κανονική αίτηση σημαίνει ότι ένας πιθανός ετών ε, άσυλο ε, έχει ξεφύγει από μια διαμάχη σε τρίτη χώρα και θέλει να ζητήσει ε, θεώρηση Σέγγεν. Δεν μπορεί να ζητήσει ανθρωπιστική θεώρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα, μπορεί όμως ε, να ζητήσει ε, διεθνή προστασία. Και το κράτος μέλος μπορεί έτσι να εξετάσει εάν θα πρέπει να εκδοθεί θεώρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα ε, ή θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύως. Ένα ετών άσυλο λοιπόν κάνει αίτηση για μια τέτοια θεώρηση, τα χαρτιά του δεν είναι εντάξει ή δεν έχει τα απαραίτητα χρήματα. Κάτι που συχνά ισχύει για ανθρώπους ε, που ε, προσπαθούν να ξεφύγουν από κάποια διαμάχη. Στην περίπτωση αυτή δεν ε, μπορεί να λάβει θεώρηση διότι δεν πληρεί τα κριτήρια ο ετών. Αλλά το 19.4 λέει ότι οι αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσει για λόγους εθνικού συμφέροντος, όχι όμως λόγω διεθνών υποχρεώσεων, όπως είδαμε στην αρχή της παρουσίασης. Ε, αν λοιπόν θεωρεί απαράδεκτη η αίτηση, Υπάρχουν εδώ δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν έχει δικαίωμα προσφυγής ο ετών, διότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον κώδικα θεωρήσεων. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι η διαδικασία για τη θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύω αναφέρει τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις ως λόγο για την έκδοση της θεώρησης αυτής, αλλά ήδη έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία αυτή ο ετών, διότι έχει θεωρηθεί απαράδεκτη η αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 19. Άλλο παράδειγμα αυτών των ασυνεπιών στον ε, ισχύοντα κώδικα Σέγγεν ε, είναι η περίπτωση ενός ασθενούς που ζητάει θεώρηση για να ε, λάβει περίθαλψη και θεραπεία σε κράτος μέλος. Ε, κάνει λοιπόν αίτηση για βίζα, υποβάλλει αίτηση για βίζα και για γιατρικούς λόγους. Μπορεί λοιπόν τα, να μην έχει τα απαραίτητα έγγραφα ή να μην έχει τα λεφτά που απαιτούνται. Μπορεί λοιπόν και εδώ να γίνει παρέκκληση για ανθρωπιστικούς λόγους ή για λόγους εθνικού συμφέροντος ε, σύμφωνα με το άρθρο 19.4. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι ε, ε, αυτή η σοβαρά ασθενής θεωρηθεί, ότι η αίτησή της θα θεωρηθεί παραδεχτή και θα γίνει η διεκπαιρέωση της αίτησής της. Οι αρχές λοιπόν ήδη θα έχουν να αναγνωρίσουν ε, τον ανθρωπιστικό λόγο για το παραδεκτό της αίτηση, αλλά αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τον ισχύοντα κώδικα θεωρήσεων. Και εάν εκδώσει ένα κράτος θεώρηση περιορισμένη εδαφική ισχύω ε, δεν είναι σαφές αν αυτή έχει εκδοθεί με βάση τον κώδικα θεωρήσεων, διότι δεν υπάρχουν εδώ σαφείς κανόνες. Και έτσι φτάνουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ελλείψεις και ασυνέπειες που ε, έχει διαπιστώσει η μελέτη. Ιδιαίτερα οι συστάσεις υπαριθμών 6, 7 και 8 προτείνουν κάποιες λύσεις. Για παράδειγμα, η σύσταση υπαριθμών 6 προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει περισσότερη συνέπεια στην ε, εφαρμογή των κανόνων, δηλαδή να προσθεθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις στον κατάλογο λόγων αποδοχής της ε, αίτησης στο άρθρο 19.4. Επιπλέον η μελέτη προτείνει στην σύσταση υπαριθμών 7 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει ο κώδικας θεωρήσεων να περιέχει σαφή διαδικασία για την υποβολή και διεκπαιρέωση αιτήσεων για την θεώρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Το σημαντικό εδώ είναι η θεώρηση ανθρωπιστικού χαρακτήρα να είναι ξεχωριστή κατηγορία θεωρήσεων και τα κράτη-μέλη να είναι υποχρεωμένα να κάνουν αξιολόγηση σύμφωνα με το 25.1 και σύμφωνα με το άρθρο 19.4. Δηλαδή να διαπιστώσουν αν είναι εάν δικαιολογείται η παρέκκληση από τους ισχύοντες κανόνες και μια τέτοια διάταξη μπορεί να διατύπωθεί με τρόπο ανάλογο με τον κανόνα που ισχύει για τις κανονικές θεωρήσεις στον κώδικα θεωρήσεων. Και επίσης έχουμε την σύσταση υπαρθμών 8 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει να υπάρχει ρητό δικαίωμα προσφυγής σε περίπτωση άρνησης έκδοσης ε, θεω, ε, θεώρησης ε, ανθρωπιστικού χαρακτήρα, καθώς και σε περιπτώσεις όπου θεωρείται απαράδεκτη η αίτηση. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο συμπέρασμα της μελέτης. Τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει μια σειρά διαφόρων καθεστώτων ε, για θεωρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, διστάζουν όμως ε, να στηρίξουν ε, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Στην σελίδα 49 της μελέτης θα βρείτε το σχετικό διάγραμμα, όπου φαίνεται ότι 16 κράτη-μέλη έχουν ή είχαν κάποιο είδος καθεστώτος ε, έκδοσης θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα, είτε αυτές ήταν εθνικές, είτε ήταν θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύω. Γενικά φαίνεται ότι ως εξαίρεση έχουν, εφαρμοστεί, έχουν εκδοθεί αυτές οι θεωρήσεις. Να σχολιάσω όμως εδώ τον χάρτη αυτόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες ε, που έχουμε, δεν είναι πάντα σαφές τι είδους θεώρηση έχει εκδώσει ένα, ένα κρατός Γι' αυτό και για να μπορούμε να έχουμε μια συνολική επισκόπηση των πρακτικών των κρατών μελών, ε, περιλαμβάνει ο χάρτης αυτός ε, και τις θεωρήσεις ε, μακράς διαρκείας ε, ε, και μικρής διαρκείας, καθώς και τις θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύω. Επειδή δεν υπάρχει ευρωπαϊκός μηχανισμός που να παρακολουθεί την έκδοση των θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη και ενιαία εικόνα σχετικά με την έκδοση αυτών των θεωρήσεων και έτσι είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πώς χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη αυτές τις θεωρήσεις. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ο αριθμός θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ε, ισχύω ε, που έχουν εκτός τα κράτη-μέλη, περίπου 300.000 ε, το 2012. Δεν γνωρίζουμε όμως τους λόγους έκδοσης αυτών των θεωρήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα ε, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν στατιστικές στην Κομισιόν σχετικά με, για παράδειγμα, τον αριθμό θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύως που εκδίδονται. Στις ε, σελίδες 14 ε, και 15 της μελέτης ε, θα βρείτε παραπομπές σε άλλες μελέτες που έχουν εκπονηθεί. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι πάνω από το μισό των κρατών μελών αναγνωρίζουν ή έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για μια θεώρηση τέτοιου είδους, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί κάτι τέτοιο για πρακτικούς λόγους όπως είναι το μοίρασμα του άχθους μεταξύ των κρατών μελών, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί κατά την εκπόνηση κανόνων Σέγγεν για τις θεωρήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έτσι φτάνω στο τι μπορεί να γίνει για να προωθήσουμε την χρήση θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Οι συστάσεις υπαριθμών 1, 2, 3 και 4 έχουν να κάνουν με κάποια από τα γενικότερα θέματα όπως είναι η διαχείριση των συνόρων και ο έλεγχος των συνόρων, ενώ η σύσταση υπαριθμών 12 σχετίζεται άμεσα με τον κώδικα θεωρήσεων. Στην ε, σύσταση αυτή ε, προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει έκκληση για έναν μηχανισμό παρακολούθησης, διότι ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να βασιστεί στον μηχανισμό κοινοποίησης που ήδη θεσπίζεται στον κώδικα θεωρήσεων, που απαιτεί από τα κράτη-μέλη να ε, συντάσσουν ετησίως στατιστικές σχετικά με τις θεωρίες περιορισμένη εδαφική ισχύω που εκδίδονται και τις αιτήσει που έχουν υποβληθεί. Ένας μηχανισμός παρακολούθησης μπορεί να διασφαλίσει και να προωθήσει πιο ενιαία εφαρμογή των κανόνων και μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση. Επιπλέον θα υπάρχει περισσότερη σαφήνεια στον κώδικα, κάτι που είναι απαραίτητο και ε, θα υπάρχει περισσότερη σαφήνεια. Έτσι θα είναι πιο σαφείς οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και είναι σαφές ότι το ζήτημα των θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται συνεχώς η συζήτηση αυτή για το αν θα πρέπει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα, ένα τέτοιο σύστημα. Και βλέπουμε τελικά ότι θα πρέπει να γίνει και μία συζήτηση μετά την παρουσίασή σας και δυστυχώς δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο αυτή τη στιγμή στη σημερινή μας συνεδρίαση θα θέλαμε πάρα πολύ πραγματικά, ιδίως όσον αφορά τα δύο βασικά σας συμπεράσματα, να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις και να γίνει μια κάποια συζήτηση. Είναι ήδη εδώ πέρα η κυρία Γκρίσμπεκ, η οποία είναι υπεύθυνη για το επόμενο ζήτημα. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να δώσω μια μάχη με τη γραμματεία η οποία τα τελευταία 15-14 λεπτά με πιέζει γιατί είχε προβλέψει πολύ σωστά ότι ε, δεν απέμενε πάρα πολύ χρόνος. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε το εξής. Ο κύριος ε, Λόπες Αγγιλάρ έχει ήδη έναν γράφο εργασίας και είπε ότι στα πλαίσια αυτού του νέου γράφου εργασίας θα έχουμε μια νέα ανταλλαγή απόψεων. Θα γίνει λοιπόν μια περαιτέρω συζήτηση. Θα θέλαμε να σωματώσουμε σε αυτή τη νέα συζήτηση και το ζήτημα των θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Η νέα λοιπόν αυτή συζήτηση θα γίνει πολύ σύντομα. Θα ενταχθεί λοιπόν και το δικό σας το ζήτημα στη μερίσια διάταξη. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο αλλά φαντάζομαι ότι η γραμματεία δεν θα μου επιτρέψει αυτή τη στιγμή να σας δώσω το λόγο. Ναταλή, θέλεις τώρα να καλύψουμε το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη. Α, κύριε Πρόεδρε, αρκεί να προβλεφθούν αυτά τα 45 λεπτά συζήτηση. Είτε μπορούμε τώρα να καλύψουμε αυτά τα 45 λεπτά, ή να το κάνουμε και αργότερα. Αρκεί να προβλεφθεί ο απαραίτητο χρόνο για να γίνει η συζήτηση για τη δική μου την έκθεση, που είναι εξίσου σημαντική με το ζήτημα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Αλλά μπορώ να παραμείνω και περισσότερο, αν θέλετε, να κάνουμε τη συζήτηση αυτή λίγο αργότερα. Βέβαια θα καθυστερήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και με τα επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Ήμπως προτιμάτε κύριε Πρόεδρε να συντομεύσουμε το χρόνο συζήτησης της δικής μου έκθεσης, πράγμα το οποίο δεν θα ήθελα να σας πω την αλήθεια. Σε ευχαριστούμε να τα λύσουν απόλυτα σαφή, σε ευχαριστούμε που μας βοήθησες τόσο πολύ. θα προτιμούσα πραγματικά οι Γάλλοι να τηρήσουν το στερότυπο το οποίο υπάρχει για αυτούς ότι γενικά δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Αν να μας βοηθάς όπως μας βοήθησες τώρα, καλύτερα να μας βοηθάτε. Λοιπόν, να είμαι λίγο πιο σαφής. Έχουμε ένα έγγραφο εργασία του κυρίου Λόπετ Αγκουιλάρ, στα πλαίσια του οποίου θα γίνει μια ουσιώδη ανταλλαγή απόψεων και στα πλαίσια τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να καλύψουμε και το ζήτημα των θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα αυτό. Εκπονήθηκε η μελέτη την οποία η Επιτροπή μα ζήτησε. Έχει καταλήξει συγκεκριμένα συμπεράσματα η μελέτη αυτή και πρέπει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Πάντως, ξέρετε ότι στο παρελθόν, όταν είχαμε κάνει μία συζήτηση για τις θεωρίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα, είχαμε μία πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση και νομίζω ότι κάτι ανάλογο θα πρέπει να γίνει και στην επόμενη συζήτηση που θα γίνει για το ζήτημα αυτό. Και ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι είχαμε τη δική σας την παρουσίαση και ότι έχουμε στα χέρια μας τη μελέτη την οποία εκπονήσατε. Και όπως σας είπα, για το έγγραφο εργασία του κυρίου Λόπες Αγκουιλάρ πρόκειται σύντομα να γίνει μια νέα συζήτηση και στα πλαίσια της συζήτησης αυτής θα συμπεριλάβουμε και το ζήτημα των θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Θα το αποφασίσουμε αυτό στη συνάντηση που θα έχουμε με τους τονιστές τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Για άλλη μια φορά, κυρία Ιμπεν Γένσεν, σας ευχαριστώ πολύ για την μελέτη σας και για την παρουσίαση που κάνετε. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο σημείο 7 τη σας διάταξη, ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου τη αθωότητο και του δικαιώματο παράσταση του κατηγορουμένου στη δίκη στο πλαίσιο ποινική διαδικασία. Σας υπενθυμίζω ότι η προτινόμενη οδηγία αποτελεί συνέχεια προηγούμενων οδηγιών από τη δέσμη οδηγιών του 2009 όσον αφορά την ενίσχυση των διαδικαστικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Έγιναν επιπλέον δύο προτάσεις, η μία αφορά τα παιδιά και τις ποινικέ διαδικασίες καθώς επίσης και τη νομική αρρωγή και Ετέθη επίση και το ζήτημα του τεκμηρίου τη αθεότητα, που αποτελεί βασικότατο δικαίωμα στα πλαίσια των σύγχρονων ποινικών διαδικασιών, στα πλαίσια δημοκρατιών που βασίζονται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα συζητήσουμε τι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί. Θα δώσω καταρχά το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Γκρίσμπεκ. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στου κοιόδη εισηγητέ. Ξεκινάμε όμω τώρα με την Άταλη Γκρίσμπεκ, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Κλώτα, αγαπητοί συνάδελφοι. θα σας καθησυχάσω, δεν θα σας ε, δημιουργήσουν προβλήματα οι Γάλλοι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη για να έχουμε, ελπίζω, για μια ακόμη φορά μια πλούσια συζήτηση για αυτό το σχέδιο οδηγίας που έχει να κάνει με την ενίσχυση, όπως λέει ο τίτλος, ε, μιας πρώτας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενίσχυση, λοιπόν, των δικαιωμάτων σε αυτό το τεκμήριο της αθότητας. Ε, πρόκειται για την τρίτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό Αρχές Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα περίπου, σας παρουσίασα το πρώτο σχέδιο έκθεσης ε, που έχει ένα πολύ γενικό στόχο, δηλαδή με 44 τροπολογίες ε, που καταθέτω να ενισχυθεί η προστασία αυτού του δικαιώματο. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, όπω ζήτησαν ορισμένοι συνάδελφοι, επιμηκύθηκε και μέχρι ε, τώρα έχουμε λάβει 180 τροπολογίε. Φυσικά και με χαροποιεί ιδιαιτέρω το ενδιαφέρον που δείχνουν οι συνάδελφοι για το θέμα αυτό, για αυτή την πολύ σημαντική αρχή του τεκμηρίου αθότητα. Και χαιρετίζω την πολύ μεγάλη συμμετοχή πολλών συναδέλφων που δείχνει πόσο σημαντική είναι η οδηγία και πόσο σημαντική είναι η αρχή. Είπε και εσύ, Κλόντ, ότι η αρχή αυτή είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Είπαμε ότι θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τα πράγματα. Είχαμε και στην 789 τη σύμβαση ως πυλώνα της προστασίας ε, δικαιωμάτων, ε, ιδίως στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, του τεκμηρίου αθότητας. Είναι πολύ σημαντικό το δικαίωμα υπεράσπισης γενικά, ιδίως ε, για εμάς, για την Ευρωπαϊκή Επικράτη, για να εγγυηθούμε στον Ευρωπαίο Πολιτό δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. να αποφύγουμε αυθαιρεσίες όσο μπορούμε, καθώς και καταχρήσεις στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών για να τα πω έτσι σφαιρικά και γρήγορα, γρήγορα, η γραμμή βασική ε, που πιστεύω ότι χαρακτηρίζει τις περισσότερες τροπολογίες και των σκιωδών που τους ε, ευχαριστώ γιατί από την αρχή των εργασιών συμμετείχαν. Τέσσερις ιδέες βασικά μπορούμε να διακρίνουμε, μεγαλύτερη νομική προστασία βέβαια. Είναι και το πνεύμα μάλιστα της πρότασης οδηγίας η ενίσχυση μία θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να ενισχύει από την πλευρά της αυτή την προσέγγιση της Κομισιόν, μια οδηγία φιλόδοξη και τέλος μια οδηγία που βέβαια, όπως και με πολλά κείμενα, θα αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων ε, προς τα πάνω και προς τα κάτω ή δυνατόν. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για τις αυτές που βελτιώνουν, συμπληρώνουν, εμπλουτίζουν το κείμενο. Δεν θα τα καλύψω διεξοδικά και εξαντλητικά. Έχω από χθε μόλις το βράδυ τη γαλλική μετάφραση των τροπολογιών. Θα περιουστώ σε 7-8 σύντομες παρατηρήσεις. Ηρεμήστε, δεν πρόκειται να σας αναπτύξω εδώ όλο το περιεχόμενο αυτών των πολλών τροπολογιών. Πρώτον λοιπόν, οι περισσότεροι συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους επιβεβαιώνουν την ανάγκη διεύνηση του πεδίου εφαρμογή όπω προτείνω και εγώ στο σχέδιο έκθεσή μου. Από τη μια πλευρά υπογραμμίζουν κάποιε τροπολέ ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν και τα νομικά πρόσωπα στο πεδίο εφαρμογή και κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο διότι και τα νομικά πρόσωπα μπορούν ε, να ε, υποβληθούν ε, μπορούν να γίνουν αντικείμενο επιβολής ποινικών κυρώσεων, παραλυσμός τύπου όπως το αποκαλούμε, Πρέπει να υπάρξει λοιπόν η συμμετοχή αυτή. Επίσης, σε ό,τι αφορά και τις διοικητικές διαδικασίες που έχουν ποινικέ επιπτώσεις, θέλουμε να περιλαμβάνονται και αυτές ε, άλλωστε προβλέπεται και από την νομολογία του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα ποινικά ζητήματα. Με διεύρυνση παιδί εφαρμογή. Άλλε τροπολογίε τώρα λένε ότι όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η οδηγία, μάλλον τονίζονται στο στο πότε, από πότε αρχεί να ισχύει και για πόσο αυτή η οδηγία. Υπάρχει με το σκέψη 17 για την απόκτηση τεκμηρίων μέσω άσκηση πέσεων καταναγκασμού να διαγραφεί ε, ζητούν τροπολογίες και φυσικά ε, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ο καταναγκασμός ε, είναι κάτι που φυσικά δεν θέλουμε να υπάρχει. Είναι καλό να το λέμε λοιπόν συγκεκριμένο. Και για το άρθρο 4 έχουμε πολλές τροπολογίες. Είναι ένα κομβικό άρθρο για το τεκμήριο αθότητας. Συγκεκριμένα, απαγόρευση ε, της πρόορης ε, ε, ομολογίας ενοχής, η δήλωση ενοχής. Το 18ο αιώνα, από το 18ο αιώνα καταπατάται κάθε μέρα αυτό το δικαίωμα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν στις τροπολογίες την απαγόρευση ε, της δήλωσης ε, ενοχής. Πριν υπάρξει απόφαση δικαστική. Επίσης προσθέθεται κάποια εχέγγυα, κάποιες εγγύησεις και ένας πολύ λεπτός τομέας όπως είναι το τεκμεαθότητας. Ε, εδώ βλέπουμε πολλές φορές να παραβιάζεται η αρχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να βρεθεί ισορροπία μεταξύ αφενός της ελευθεροτυπίας βέβαια, αλλά και αφετέρου της προστασίας των πολιτών. για όσα θεωρούν σημαντικά. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση και χαίρομαι πάρα πολύ που κατατέθησαν τόσες τροπολογίες για αυτά τα πολύ λεπτά ζητήματα που πρέπει όμως να τα επισημάνουμε ξεκάθαρα. Τέταρτο σημείο, σύντομα. Πολλές τροπολογίες συμφωνούν με την ιδέα της συμπερίληψης σε ένα νομικό κείμενο για ποινικά ζητήματα ε, της αρχής της αναστροφής του βάρους απόδειξης. Επικίνδυνο. Αν ισχύσει. Αυτή η απαγόρευση της περίληψης λοιπόν ε, ε, που επιβεβαιώνει και η νομολογία σε πολλέ περιπτώσει. Πέμπτο σημείο. Άλλε τροπολογίε συμπληρώνουν ή διευκρινίζουν τα άρθρα 6 και 7 που αφορούν ε, το δικαίωμα ε, στη σιωπή. Πολύ καινοτόμα νεοτεριστική πρόταση στο σχέδιο οδηγίας της Κομισιόν. Δηλαδή να μην αυτοκατηγορηθεί κάποιος ή αυτοενοχοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Με όλα αυτά τα στοιχεία Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό κείμενο ε, με ισχυρή διατύπωση για τα άρθρα 6 και 7. τώρα σε ένα πολύ προσφυλές για μένα θέμα που είναι και στο επίκεντρο του σύντομα αυτού κειμένου. Συγκεκριμένα πρόκειται για το πρόβλημα των αποδείξεων που ε, αποσπώνται με παραβίαση του άρθρου περί μια φτωχοενοχοποίηση και κατάρριση του δικαιώματο στη σιωπή που είναι αναφέρει το δικαίωμα. Και εδώ έχουμε πολλέ τροπολογίε από τις οποίες ε, φαίνεται ότι συμφωνούν ε, οι συνάδελφοι, οι σκιώδες και αυτό συνιστά επίσης μεγάλη πρόοδο. Ολοκληρώνω σχεδόν κάποιες τροπολογίες εισάγουν πολύ ενδιαφέροντα νέα στοιχεία, καινοτόμα στοιχεία στην οδηγία. Και συγκεκριμένα στην παρουσίαση του ε, κατηγορούμενου ή υπόπτου ε, στην ε, κροματική διαδικασία. Αυτό και άλλα στοιχεία είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί μπορούν να βοηθήσουν στον εξυγχρονισμό των ποινικών διαδικασιών. Ελπίζω να τα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Δεν είναι βέβαια μανιχαϊστική η... η έκθεση. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και κάποια μίσθων των εγγυήσεων ε, για τους ε, υπόπτες. Υπάρχουν κάποια θέματα που ε, θα με δυσκολέψουν να τα δεχθώ, αλλά είμαι στη διάθεση όλων όσων συνέταξαν ανθρωπολογίες για να βρούμε μια βάση συνεννόησης. Θα προσπαθήσω επίσης να σας προτείνω μια πρώτη δέσμη συμβιβαστικών τροπολογιών την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολλές τροπολογίες, προσπαθώ να συμφιλιώσω τις διαφορετικές απόψεις. Ίσως αυτό να είναι πολύπλοκο εγχείρημα, ενίοτε, αλλά αυτό είναι ε, δουλειά που πρέπει να γίνει. Στόχος είναι να βρούμε κάποιες κοινέ γραμμές για να είμαστε έτοιμοι πριν τους τριμμένους διαλόγου. Είναι σημαντική η πρόταση αυτή. Ακόμη πιο πολύ δε, καθότι σήμερα στην Ένωση και με τις επαφές που είχα βλέπω ότι βλέπουμε ένα είδος διάβρωσης της αρχής του τεκμηρίου αθότητας. Άρα αυτό το σχέδιο οδηγίας νομίζω ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε αυτή τη σύντομη έκθεση. Δεν θα είναι δηλαδή η έκθεση τόσο μακροσκελής όσο ήταν η σημερινή μου παρουσίαση. Και ελπίζω να ανταποκριθεί στι φιλοδοξίες και προσδοκίε του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, ελπίζω ότι δεν μακρηγόρησε. Δέκα λεπτά, ε, εντάξει, καλά τα πήγα. Ούτε καν δέκα. Uh, Μα Μιλήσατε λοιπόν για το τεκμήριο για το δικαίωμα παράσταση. Δύο πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Δεν καλύψατε τόσο πολύ χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάταλ. Είναι παρόντε όλοι οι σκιώδει συζητητέ. Επομένω, μπορούμε να έχουμε πλέον μια καλή συζήτηση. Καταρχά, η κυρία Γκάλαπ για το ΕΛΚ δεν είναι παρούσα. Η κυρία Μόσκα θα πάρει το λόγο για την εκπροσωπήση εξ ονόματο του Ελκ παρακαλώ. Η κυρία Μόσκα είναι εδώ στην αίθουσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, προσωπώντος την κυρία Κιγκαγκάλη, η οποία είναι σκιώδη συγγήτρια για το ΕΛΚΑ. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσω το μήνυμα το οποίο θέλει να αποστείλει. Καταρχάς σας ζητά συγγνώμη, έπρεπε να είναι σε συνεδρίαση του Προεδρείου, επομένως δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα σας διαβάσω λοιπόν το κείμενο το οποίο μου έδωσε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για την εργασία που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμή. Ο τελικό στόχο τη συλλογική μα προσπάθεια είναι να εγγυηθούμε δίκαιε δίκαιε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων υπεράσπισης όπως εμπεριέχονται συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χάρτη θεμελιώδων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις αλλαγές που έχει προτείνει η συγκήτρια όσον αφορά την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε στόχο να επιτευχθεί ένας γενικότερος στόχος προστασίας υποπτών κατηγορουμένων σε ποινικέ διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπερβούμε τα όσα προβλέπονται για τα δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων σε σημείο δηλαδή που θα θέτουμε να αμφιβόλου την ένωμη τάξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση προκειμένου από τη μια να τηρείται το δικαίωμα τεκμηρίου αθεότητος και δικαίωμα παράστασης και από την άλλη όμως θα πρέπει να τηρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις στα πλαίσια μιας ποινική διαδικασίας. Θα πρέπει επίσης να σεβαστούμε τα εθνικά νομικά συστήματα των κρατών μελών και θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε μια αποτελεσματική, πιο αποτελεσματική ποινική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε το δικαίωμα σιωπή που αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και από την άλλη όμως θα πρέπει ο ύποπτος κατηγορούμενος να συνεργάζεται σωστά στα πλαίσια της ποινική διαδικασίας. Είναι ευθύνη μας να καταφέρουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων και την... χωρίς όμως να βάλουμε κατά της αρμονικής διεξαγωγής διαδικασίας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας και θα πρέπει να συμβάλλουμε βέβαια και στην αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη συμφωνούμε σε πάρα πολλά σημεία με την εισηγήτρια, όπως για παράδειγμα το ότι θα πρέπει η οδηγία αυτή να περιέχει μία αναφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά επίσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Πολιτικών Δικαιωμάτων, καθώς επίσης και στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συμφωνούμε επίσης ότι το βάρος απόδειξης θα πρέπει να παραμένει στα πλαίσια της εισαγγελικής αρχής, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μόνο δίκαιες δίκες και οποιαδήποτε αμφιβολία θα πρέπει να είναι υπέρ του κατηγορουμένου στα πλαίσια της ποινική διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία κατηγορουμένου υπόπτου σε σχέση με πληροφορίες οι οποίες διαραίουν προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτό δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ενισχυμένη προστασία για τον ύποπτο και τον κατηγορούμενο. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια που κάνει η συγγήτρια να καταλήξει σε συμβαστικές τροπολογίες και θα ήθελα και εγώ σκιώδη συγγήτρια να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ ο Πρόεδρος, μας είπατε ποια είναι η άποψη της κυρίας Γκάλ, εξ τώρα των Σοσιαλιστών η κυρία Μπίργκιτ Σίπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σχεδόν ότι η πρόταση της Επιτροπής περιέχει πολύ λίγα συγκεκριμένα πράγματα και στην πράξη το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα παράστασης ε, στη δίκη ε, στην πράξη πρέπει να ενισχυθούν αλλά δεν περιέχονται εδώ συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, συμφωνώ με την Νάταλη Κρίσπεκ που στην ε, έκθεσή της ε, με τις ε, τροπολογίες έχει επισημάνει κάποια από τα σημεία αυτά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί της. Θα πρέπει το τεκμήριο αθωότητας να ισχύει χωρίς εξαιρέσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καταναγκασμός και δεν θα πρέπει να ε, επιτρέπεται καμία παραβίαση αυτών των αρχών. Θεωρώ τις τροπολογίες μου προσθήκη στις εργασίες ε, της εισηγήτριας. Θα ήθελα να έχω καθορισμό της ε, προθεσμίας θα πρέπει το κλείσιμο της διαδικασίας να ισοδυναμεί με ε, απόλυτο ξεκαθάρισμα του θέματος ε, της αθωότητας. Το τεκμήριο αθωότητας εκτός των δικαστηρίων με ε, άτυπη ε, διαβίβαση πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, δεν προστατεύεται. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πώς παρουσιάζεται ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο. Δηλαδή, ε, οι χειροπέδες ε, ή άλλα τέτοια μέτρα δεν επιτρέπεται ε, να έχουν ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί ήδη ένοχος. Θα πρέπει και εκτός των δικαστηρίων ε, να προστατεύει το τεκμήριο αθωότητας, κάτι που δεν σημαίνει αυτή τη στιγμή. Επίσης, ο κατηγορούμενος δεν ε, θα πρέπει να έχει μειονεκτήματα ε, επειδή βραχυπρόθεσμα, αλλά χωρίς δικό του φταίξιμο δεν μπορεί να παρευρεθεί σε ποινική διαδικασία. Γι' αυτό είναι σημαντικό η, η συγγήτρια να αναφερθεί στα δικαιώματα του καθενός, διότι μόνο αν γνωρίζει κανείς τα δικαιώματα μπορεί να διασφαλίσει τον σεβασμό τους. Ε, πιστεύω ότι θα βρούμε καλούς συμβιβασμούς ε, μαζί με την εισηγήτρια. Σε αντίθεση με την πρόταση της Κομισιόν, θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στελιόν για την ομάδα Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Η ομάδα μας ε, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την έκθεση αυτή ήδη έχει πει ότι η έκθεση της κυρίας Κρίσπεκ αποτελεί εξαιρετική βάση για συζήτηση. Ίσως ε, γι' αυτό να έχουμε κάπως λιγότερες τροπολογίες από πλευράς της ομάδας μας. Ε, δεν οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος ο μικρός αριθμός τους, ε, οφείλεται στην εξαιρετική ποιότητα της έκθεσης. Η συγγήτρια είπε ότι θα παρουσιάσει σύντομα συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, στην περίπτωση αυτή, εγώ θα προσπαθήσω μόνο να πετύχω βελτιώσεις όπως προτίθηκαν από τους Πρασίνους και την ομάδα SND για να συμπληρώσουμε τη δουλειά που ήδη έχει γίνει. Δεν ε, θα υποστηρίξω όμως καμιά συμβαστική τροπολογία που θα υπονομεύσει το επίπεδο της έκθεσης αυτής. Ε, μπορώ να είμαι σύντομος. Ε, μία παρατήρηση έχω επί της ουσίας που πιστεύω ότι είναι σημαντική προσθήκη σε αυτά που ήδη συζητήσαμε. Αναφέρομαι στο τι στοιχεία μπορεί να λάβει υπόψη του ο δικαστή ε, ω ελαφρυντικά στοιχεία. Μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει υπόψη του την ενεργό συμμετοχή ε, του κατηγορούμενου στην ποινική διαδικασία. Αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στι τροπολογίε τη κυρία Κρίσπεκ και πιστεύω ότι μπορεί να συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ. Εξαιρετικό ο έπαινος που ακούτε για την έκθεσή σας από τους Πρασίνους, ο κύριος Άλπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Κρίσπεκ, για αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόκληση θα είναι να καταφέρουμε να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη στα πρότυπα που θέλουμε εμείς να πετύχουμε και που θα θέλαμε να θεσπιστούν ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την προστασία των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Η κυρία Σίπελ ε, ήδη είπε ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε στο βαθμό που είναι δυνατή την μεταφορά του βάρους αποδείξεως. Δεν ε, θα πρέπει να περιοριστούν τα δικαιώματα και θα πρέπει να υπάρχουν και αυστηροί κανόνες σχετικά με το παραδεκτό των αποδείξεων. Οτιδήποτε είναι αποτέλεσμα καταναγκασμού θα πρέπει να αποκλείεται. Θα πρέπει αυτό να θεσπίζεται γραπτός, ε, το είπε ήδη και η συγγήτρια. θα μπορέσουμε τότε να δούμε σε τι βαθμό θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στο Συμβούλιο. Πάντως είμαι πολύ αισιόδοξο. Πιστεύω ότι εδώ θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εξαιρετική έκθεση της κυρίας Γκρίσμπεκ. Μια έκθεση με την οποία συμφωνούμε απόλυτα. Οι τροπολογίες που έχει καταθέσει κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Με αυτή δηλαδή που μας είχε παρουσιάσει στα πλαίσια της εκθεσής της. Κάποιες παρατηρήσεις μόνο να κάνω σε σχέση με τις τροπολογίες που εγώ κατέθεσα. Όσον αφορά το ζήτημα της ε, αντιστροφής του βάρους απόδειξης. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η δυνατότητα αντιστροφής του βάρους απόδειξης. Και μάλιστα, εγώ είχα αναφερθεί και στην ε, τήρηση της ε, αρχής να μπορεί να αντιταχθεί κανείς στις αποδείξεις που κατατίθενται. Δηλαδή, η απόδειξη να προβλέπεται τόσο για την υπεράσπιση όσο και για την, τον φορέα της κατηγορίας. Θα πρέπει δηλαδή να μπορεί και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο ίδιος ο ύποπτος να παρέχει τις δικές του αποδείξεις. Τώρα, όσον αφορά τις αναφορές που γίνονται για τον ύποπτο και τον κατηγορούμενο και όσον αφορά τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται σαν να έχει ήδη καταδικαστεί ο άνθρωπος αυτός. Θα πρέπει να επεκτείνουμε ακόμα και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την αρχή αυτή της απαγόρευσης των πρόωρων δηλώσεων ε, ενοχής. Θα πρέπει δηλαδή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως σε κάποιες συνεντεύξεις ε, ή σε κάποια ρεπορτάζ τα οποία κάνουν κατά τη διάρκεια μιας ποινική διαδικασίας, να μην αναφέρονται σε αυτόν ως ε, ήδη ένοχο, αλλά απλώς ως ύποπτο ή κατηγορούμενο. Τώρα, όσον αφορά επίση το δικαίωμα σιωπή. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα σιωπής ε, ως ε, καταδικαστική απόδειξη ή ότι θα μπορεί να αποτελέσει ποτέ τεκμήριο καταδίκης και νομίζω ότι θα πρέπει να απογορευτεί και οποιοδήποτε καταναγκασμό για την απόσπαση αποδεικτικών στοιχείων. Δεν θα πρέπει να προβλέπεται καμία απολύτω απόκληση, εξαίρεση όσον αφορά του μηχανισμού καταναγκασμών. Γιατί διαφορετικά νομίζω θα καταλήξουμε πραγματικά σε βασανιστήρια. Τώρα, όσον αφορά την δυνατότητα μη συνεργασίας, θα ήμουν κάπως πιο προσεκτική όσον αφορά την θέσπιση αυτής της αρχής αυτού του δικαιώματος, διότι ε, φοβάμαι ότι ενδεχομένω εδώ πέρα ελοχεύει ένας κίνδυνος παρερμηνίας του δικαιώματος αυτού. γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές ε, η ε, αρχή της μη συνεργασίας, εφόσον εφαρμοστεί όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή στο κείμενο, ενδεχομένως να μην λειτουργήσει υπέρ της ποινική διαδικασίας. Όσον αφορά τώρα το άρθρο 8, προφανώς χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον κατηγορούμενο ιδίω κατά τη διάρκεια τη ποινική διαδικασία ει βάρο του. Θα πρέπει δηλαδή ο άνθρωπο αυτό να ενημερώνεται καλύτερα, να υπάρχει καλύτερη γνωστοποίηση τη νομοθεσία που τον αφορά. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος να γνωρίζει ακριβώς πώς διεξάγεται η ακροματική διαδικασία και ποια είναι η ε, νομοθεσία η οποία τον αφορά. Και θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός βέβαια να μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν έμπιστο δικηγόρο ή τουλάχιστον να έχει πρόσβαση σε έναν δικηγόρο ο οποίος θα ανατεθεί σε αυτόν από την δικαστική αρχή. Επίσης αναφερόμαστε στην ε, δυνατότητα να ανοίξει πάλι η δίκη σε περίπτωση που δούμε ότι υπάρχουν νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να θέσουν ένα αμφιβόλο την δικαστική απόφαση που ήδη έχει λεφθεί, ιδίω όταν πρόκειται για καταδικαστική απόφαση. Δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα σε δεδικασμένο, σε νεμπίση NIDEM, αλλά στη δυνατότητα να επανεξεταστούν κάποια νέα αποδεικτικά στοιχεία στα πλαίσια μια νέα δικαστική ε, διαδικασία. Όπω ακριβώ γίνεται σε περίπτωση δικαστικού σφάλματο. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο κατηγορούμενο, ακόμα και αυτό ο οποίο έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση να μπορεί εκ νέου να έχει τη δυνατότητα μια νέα δίκη. Σε περίπτωση δικαστικού επίσης θα πρέπει ο κατηγορούμενο, ο καταδικαστή ουσιαστικά, να έχει πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή αποζημίωση. Βέβαια, η οικονομική αποζημίωση από μόνη της δεν νομίζω ότι μπορεί να αποκαταστήσει την ηθική κοινωνική ζημία την οποία υφίσταται ο καταδικασμένος, το γεγονός ότι έχει στερηθεί όλες τις ελευθερίες τις οποίες είχε στο παρελθόν και μία παρατήρηση όσον αφορά την εφαρμογή της ίδιας οδηγίας. Νομίζω θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία αυτή μέχρι το τέλος της δικαστικής ποινική διαδικασίας και ότι η δικαστική αυτή διαδικασία ξεκινά από την πρώτη στιγμή που θα έχουμε την παραμικρή κατηγορία κατά του υπόπτου ή του κατηγορούμενου. Νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει η οδηγία αυτή να καλύπτει και τις τρεις φάσεις της ποινική διαδικασίας και να μην ισχύει μόνο στα πλαίσια της τελευταίας φάσης, όταν δηλαδή καταλήγουμε συνήθως σε μία οριστική απόφαση. Επίσης, όσον αφορά το ζήτημα των προσωπικών ελευθεριών, κάποια προσωπικά δεδομένα, όσον αφορά το DNA, κάποια, κάποια άλλη βιολογική δείκτηση, κάποια άλλα βιολογικά δεδομένα. Νομίζω ότι ε, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μέσα αυτά μόνο όταν κρίνεται πραγματικά αναγκαίο και όταν ε, το ζητήσει αυτό η ε, επίσημα εισαγγελία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι παίρνουν το λόγο όντω δικηγόροι, νομομαθείς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητές οι οποίοι έχουν εμπεριστατωμένες γνώσεις στον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ να είστε λίγο πιο ευσύνοπτοι στις παρεμβάσεις. Η κυρία Ντατή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Ανταλή Κρίσπε και την εργασία που έχει επιτελέσει και για όλες τις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεσή της. Ξέρω ότι συνεργάστηκε πολύ καλά με τον Σκιώδη συγητή, με τη Σκιώδη μάλλον συγήτρια, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, την κυρία Κιν Καγκάλ, αλλά συνεργάστηκε πολύ αποτελεσματικά και με τους υπόλοιπου κιόδη εισηγητή και βλέπουμε ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, μια πολύ καλή συμβαστική λύση όσον αφορά την έκθεση αυτή. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μια νομοθετική δέσμη που περιέχει πρόταση οδηγίες όσον αφορά επίσης και το ευεργέτημα παινίας, την δικαστική αρρωγή. Εγώ είμαι εισηγήτρια για το ζήτημα αυτό και στα πλαίσια της δέσμης αυτής μέτρων ξέρετε ότι υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στα διάφορα νομοθετικά κείμενα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνέπεια. Προκειμένου να έχει κανείς λοιπόν το ευεργέτημα παινίας θα πρέπει μάλλον να έχει πρόσβαση στο ευεργέτημα παινίας προκειμένου να καταφέρει επίσης να προασπίσει και το δικαίωμα του τεκμηρίου αθότητος Και θα πρέπει βέβαια να έχει κανείς πρόσβαση στην αρχή αυτή προτού καταδικαστεί κανείς όσον αφορά το τεκμήριο αθωότητας και όσον αφορά το δικαίωμα παράστασης, ε, Ω προ τι δύο αυτέ αρχέ, πραγματικά θα κρυθεί η δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τη. Και πρέπει επίση να δούμε και ποιο είναι το προσωρινό πεδίο εφαρμογή. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση να παρατεθεί το δικαίωμα αυτό όσον αφορά το τεκμήριο αθότητα σε όλα τα στάδια της διαδικασία, όπως υπόθηκε μέχρι την τελική απόφαση όπως μόλις τώρα το είπε και η κυρία Φεράρα. Όσον αφορά βέβαια του κατηγορουμένου και του υπόπτου, θα πρέπει να χαίρουν όλων των δικαιωμάτων στα πλαίσια τη ποινική διαδικασία. Διαφορετικά, πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένω να διηγηθούμε σε μια εναρμόνιση προ τα κάτω, σε μια ισοπαίδωση σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν καταλήξουμε δηλαδή σε ελάχιστα πρότυπα. Επίση, θα πρέπει να γίνει μια σαφή αναφορά στο ότι θα πρέπει να προστατεύουμε του ανήλικου, δηλαδή θα πρέπει στα πλαίσια της ποινική διαδικασίας να υπάρχουν συγκεκριμένε διατάξεις που εφαρμόζονται για τα παιδιά και τους ανήλικους. Στηρίζω επίσης τις τροπολογίες των συναδέλφων όσον αφορά το ζήτημα της όσον αφορά συγκεκριμένα το ευεργέτημα παινίας, όπου λέγεται ότι το ευεργέτημα παινίας θα πρέπει να εφαρμόζεται ακόμα και στους ανηλίκους. Ο επόμενος η κυρία Κινίτσι, η οποία ήταν η συζήτητρια για το θέμα που αφορά τα παιδιά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω και εγώ τη συνάδελφο Γκρίσπεκ, η οποία έκανε μια πάρα πολύ καλή εργασία όσον αφορά την οδηγία αυτή. Βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές τροπολογίες, πάρα πολλές μάλιστα, που καταδεικνύουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτή την οδηγία. και όπως ακούσαμε όντως εντάσσεται στη δέσμη αυτή μέτρων στον οδικό χάρτη που περιλαμβάνει και την οδηγία για τους ανήλικους για την οποία εγώ είμαι εισηγήτρια. Η οδηγία λοιπόν αυτή για τους ανήλικους είναι μια οδηγία που βρίσκεται σε μια πιο προχωρημένη φάση. Ήδη χθε ξεκίνησε ο τριμερής διάλογος Προσπαθούμε λοιπόν να κινηθούμε αρκετά γρήγορα για την έγκριση της οδηγίας αυτής. Ακριβώς επειδή όλοι συνειδητοποιούμε ότι η οδηγία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Να ευχαριστήσω και την ε, προλαλήσασα, δυστυχώς δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα ονόματα, η οποία αναφέρθηκε στην δυνατότητα ευεργετήματος παινίας ακόμα και στις ποινικέ εκείνες διαδικασίες που βαρύνουν ε, παιδιά και ανήλικους. Όσον αφορά τώρα την ε, οδηγία που εξετάζουμε σήμερα, θεωρώ πραγματικά ότι η κυρία Γκρίσπεκ έχει επιτελέσει μια πολύ σημαντική εργασία, καθώς επίσης και οι σκιώδεις εισηγητές φάνηκε και από τη σημερινή συζήτηση ότι όντως έχουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Θέλουμε και εδώ πέρα, όπως και στην οδηγία για τους ανήλικους, να ενισχύσουμε τις διατάξεις που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε συγκεκριμένα τα δικονομικά δικαιώματα, ακριβώς αυτό τόνισε και η δική μου πολιτική ομάδα. Γι' αυτό τόνισα και εγώ μέσω των δικών μου των τροπολογιών. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό κύριε Πρόεδρε, θέλω να αφήσω χρόνο και στους υπόλοιπους συναδέλφους να αναφερθώ σε δύο άρθρα, το 6 και το 7. Στο άρθρο 6 νομίζω ότι είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε με απόλυτη σαφήνεια το δικαίωμα της μη αυτοναχοποίησης. Όσον αφορά το δικαίωμα της σιωπής επίσης, μέσω πάλι τροπολογιών ενισχύεται το δικαίωμα αυτό. Σε καμία περίπτωση η χρησιμοποίηση του δικαίωματος, του δικαιώματος ιοπής δεν θα μπορέσει να οδηγήσει σε περιοριστικά μέτρα πριν την καταδικαστική απόφαση. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πράξη. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ατύπως ή ακατάλληλα διάφορα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να ασκηθεί πίεση στον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο προκειμένου αυτό στη συνέχεια να συνεργαστεί. Έχουμε λοιπόν υποβάλει προς αυτό αυτό κάποιες τροπολογίες. Να αναφερθώ επίσης στο δικαίωμα της σιωπής. Νομίζω ότι θα πρέπει προφανώς να ενισχυθεί το δικαίωμα αυτό. Το δικαίωμα θα πρέπει να αναγνωριστεί ακόμα και για τα άτομα εκείνα τα οποία δεν έχουν ε, χαρακτηριστεί ως ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, αλλά ακόμα και για τα άτομα εκείνα τα οποία ενδεχομένως μέσω μαρτυριών του θα μπορούσαν στη συνέχεια να ενοχοποιηθούν. Όσον αφορά το άρθρο 6, θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε αποδεικτικά στοιχεία και αν θα πρέπει να προβλέπονται άλλες μέθοδοι πέρα από τις μεθόδους καταναγκασμού προκειμένου να έχουμε απόσπαση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων. Προσπαθήσαμε και εμείς να συμβάλλουμε λοιπόν με τροπολογίες και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό κείμενο το οποίο γρήγορα ελπίζω ότι θα εγκριθεί και θα πάρει όντως τη μορφή επίσημης οδηγίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών με τους δύο τελευταίους ε, Λόπεθ Αγγιλάρ και Χολμάγερ. Φερνάντο, Χαν Φερνάντο είσαι ο πρώτο τελευταίος. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί συμφωνώ ε, με την υποστήριξη που εξέφρασαν τόσο πολλοί συνάδελφοι προς το έργο της εισηγήτρας της κυρίας Γκρισπέκ και μίλησαν για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό που αποσκοπεί την ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα για να έχουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο ποινική δικαιοσύνη. Όμω και ένα ζήτημα, ίσω το πιο λεπτό ζήτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό θα αναφερθώ, είναι η δίκη ερήμην, judgment in absentia. Όλα αυτά τα περί σιωπής, μη συνεργασίας, ε, τεκμηραθότητα, ε, φυσικά να μην γίνονται δεκτά και τα αποδεκτικά στοιχεία τα οποία αποσπάστηκαν είτε με ξαναγκασμό είτε με άλλες διαδικασίες παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν υπάρχει καμία αντίρρηση φυσικά και θα στηρίξουμε τις προτάσεις και όλοι μας θα το κάνουμε αυτό αλλά σε ό,τι αφορά την καταδίκη ερήμην τη δίκη ερήμην Υπάρχουν διαφορετικές ε, παραδόσεις στην ενόμη τάξη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά, αφορά την ε, ερημοδικία. Όπου σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατό να κρίνεται και να καταδικάζεται ένα άτομο ερήμην αν δεν συνεργάστηκε και αν με κάθε τρόπο απέφυγε παρέκαμψε την υποχρεωτική του συνεργασία με το δικαστικό σύστημα, προσπάθησε να διαφύγει να παρακάμψει το δικαστικό σύστημα. Και αυτό θεωρείται λόγος βάσιμος. Δεν είναι λάθος να στο θέμα αυτό, αλλά μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν διαφορές. Και οι υπόθεση φωτίζονται πολλές φορές από το ΔΕΚΕ, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενίοτε. Άρα είναι πολύ καλή η ευκαιρία που έχουμε να διαφωτίσουμε και εμείς την πολύ σκοτεινή αυτή σελίδα της εργασία των κρατών μελών. Για την ε, επίτευξη των στόχων για ένα χώρο ποινική δικαιοσύνη και για ενίσχυση όχι μόνο τη συνεργασία, αλλά κυρίω του να δοθεί περιεχόμενο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων των δικαστηρίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό το θέμα. Πρέπει να μας απασχολήσει και ελπίζω στα τελικά πορίσματα να περιλαμβάνονται στοιχεία που θα βοηθήσουν να υπερπαιδηθούν τα λίγα εμπόδια που υπάρχουν ακόμα μεταξύ των κρατών μελών και τις νομικές τους διατάξεις. Πρόεδρος, σε ευχαριστώ κύριε Φερνάντου, κυρία Χολμάγερ, τελευταία ομιλήτρια. Καταρχάς ευχαριστώ θερμά και την εισηγήτρια. Σημαντικά θεωρώ τα εξής όταν ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε διάφορα κράτη-μέλη έχουμε δει προβληματικές εξελίξεις. Εν μέρει αυτό οφείλεται στις εισαγγελίες, ή σε συνεργάτες ε, των αρχών που κάνουν τις έρευνες ή ακόμα και από τους δικηγόρους. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήδη ε, προδικάζεται το αποτέλεσμα. Δίδεται μια συγκεκριμένη εικόνα στο κοινό, κάτι που βρίσκω ότι είναι πολύ προβληματικό και που έχουμε δει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Έχω μακρά πείρα στο θέμα αυτό, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι υποθέσεις να εξετάζονται με βάση τα υπάρχοντα τεκμήρια και όχι με βάση την εικόνα που δίδεται στο κοινό. στην ε, οδηγία αυτό. Θα, στην οδηγία αυτή θα θέλαμε να προβλέπετε κάτι παρόμοιο σε περιπτώσεις ε, παιδιών. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητη μια τέτοια επισήμανση, αλλά θα πρέπει για όλες τις ηλικίε να ισχύει το ίδιο τεκμήριο αθότητας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Κρίσπεκ Πιστεύω ότι θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια σημεία τα οποία δημιουργούν δυσκολίες κατά τις ποινικέ διαδικασίες σε διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μόνικα. Νάταλη, ακούσαμε πολλούς επένους για το κείμενό σου. Η Κομισιόν 30 δευτερόλεπτα για να επαναλάβετε τον έπαινο. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε 30 δευτερόλεπτα και η Κομισιόν επικροτεί την ε, έκθεση της κυρίας Γκρίσπεκ και την πρόθεσή της ε, να προχωρήσει πέρα από την πρότασή μας ε, σε κάποιες πτυχές. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, διότι το τεκμήριο αθωότητας είναι ο κεντρικός πυλώνας για μια δίκαιη δίκη και θα πρέπει να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας. Επίσης επικροτούμε το ενδιαφέρον των σχεδόν εισηγητών και άλλων μελών της Επιτροπής σας στο θέμα αυτό, κάτι που έχει οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό τροπολογιών. Έχουν θυχθεί αρκετά σημαντικά θέματα στην έκθεση και στις τροπολογίες, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό προσβλέπουμε στη, στον τριμερή διάλογο που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει σύντομα και η Κομισιόν θα συνεργαστεί επικοδομητικά για να ε, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. 36 δευτερόλεπτα. Ε, ναι, μετράμε τα δευτερόλεπτα της Επιτροπής. Να, ε, σας ευχαριστώ πολύ. Νάταλη, 31 Μαρτίου θα γίνει ψηφοφορία. Θέλεις ε, να συνοψίσεις, έχεις κάτι να πεις πριν κλείσουμε. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, φυσικά τους και όλους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω σημείωσει πάρα πολλά πράγματα και για τα όσα είναι συναντικά σημεία και μπορώ να τις περιλάβω σε συμβαστικές τροπολογίες. Και όπως είπε η Ρασίντα Ντατή Γάλλο, συνάδελφος και πρώην και ε, υπουργός δικαιοσύνης ε, και ο Γιάνν Άλμπρεχτ, ε, σίγουρα πρέπει να έχουμε μια στέρεη βάση για να πάμε στον τριμερή διάλογο. Τα σημείωσα, σίγουρα δεν είχαμε πολύ χρόνο. Θα τα περιλάβω όσο μπορώ στην, ε, στη συμβασία τροπολής. Δεν ξέρω, μήπως μου δίνετε κάποια λεπτά παραπάνω να μιλήσω ή... Γιατί ε, η γραμματεία δεν θέλει να σας δώσω, αλλά θα σας δώσω εγώ δύο-τρία λεπτά, λέει ο πρόεδρος. Please go ahead while Μάλιστα. Γρήγορα, γρήγορα. Για αυτά όσα είπε η Γκάλ, διαστόματος Μποσκόρ βέβαια. Φυσικά η γενική γραμμή, το επιβεβαίωσε και η Μόνικα, είναι να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της ε, αρχής αυτής, του σεβασμού της αρχής και της προστασίας ε, των δικαιώματων. Αφήνως και των αναφορών ε, στο χάρτη, στη σύμβαση κτλ. Φυσικά και συμφωνούμε λοιπόν. Όλος ιδιαίτερος με ευχαρίστησαν τα πολύ αναλυτικά λόγια της ε, συναδέλφου Birgit Σίπελ που γνωρίζει πολύ καλά το ποινικό δίκαιο. Θα συνεχιστεί η δουλειά και σε ό,τι αφορά τις διαρροές στον τύπο Πόσο λεπτό είναι το θέμα αυτό. Πολλέ φορές έχουμε διαρροές και από τις αίθουσε των δικαστηρίων ή από το δικαστικό χώρο. Είναι λεπτό θέμα, πολλά συγκεκριμένα στοιχεία. Θα κάνουμε προτάσεις. Σε ό,τι αφορά το όσα είπε ο Ντένι Ντε σημείωσα τι παρατηρήσεις του και χαίρομαι που σε αδρές γραμμέ φαίνεται να ε, συμφωνεί το κείμενο κατά αυτόν με τι αρχέ τι οποίε υπερασπίζεται. Επίσης, η στάση, ε, το αν κάποιος είναι συνεργάσιμος, ο ύποπτος είναι συνεργάσιμος, λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας, άρα μπορώ να σας καθησυχάσω. Ε, για τον Γιάννα Άλμπρεχτ, η πρόκληση, συμφωνώ μαζί σου, είναι για να συζητήσουμε τα κράτη-μέλη και να τα πείσουμε να ακολουθήσουν ε, τη δική μας θέση. Με την κυρία Φεράρα. Επίσης συμφωνώ όπως και με την πρόταση που έκανε το τέλος ε, της απόφασης να συμπίπτει με την εκφώνηση της τιμιγορίας. Και πρώτον και κάτι άλλο κύριε Φεράρα. Να ξεκινά μια νέα διαδικασία όταν προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα το συμπεριλάβω στις συμβασικές τροπολογίες. Η Ρασίντα Ντατή που κάνει πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά ως κοιόδης είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όλοι συμφωνούμε, αλλά πρέπει να το περάσουμε και προς τα έξω, σε ό,τι αφορά την ιδιαιρότητα και το ευάλωτον των παιδιών και των ανηλίκων. Πολύ σημαντικό θέμα. Το συζητάμε και στο Intergroup για τα δικαιώματα των παιδιών, για την Κατερίνα Κινίτσι, δικαίωμα σιωπής και δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης. πρέπει να εγγυηθούμε την προστασία αυτή και για τους ε, ανθρώπους που ακόμη δεν είναι υποπτικοί σε ό,τι αφορά το άρθρο 6. Θα πρέπει να το επεξεργαστούμε εκ νέου για να διευκρινίσουμε καλύτερα το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποια στοιχεία τα οποία αποσπάστηκαν ε, δια καταναγκασμού. Θα ολοκληρώσω και είχα πολλά ακόμη να πω, αλλά θα ολοκληρώσω υπογραμμίζοντας ένα σημείο που έθεσε ο συνάδελφος Λόπεθ Αγίλα, που και αυτός γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά. Ακριβώς η ερημοδικία είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Είπε ότι κάποιες φορές το χρησιμοποιούν ως στρατηγική προστασία σε ορισμένοι υποπτή και προσπαθούν να παρακάμψουν τη δικαιοσύνη, τη δίκη. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο το γνωρίζουμε. Και για τις ερήμινα αποφάσεις. Έχουμε πολύ μεγάλη νομολογία. Κατά είναι μεγάλες οι Πρέπει ε, ο ύποπτος ή το άτομο τέλο πάντων να είναι παρόν ή να εκπροσωπείται. Αλλιώ να απαγορεύεται η έκδοση ερήμην αποφάσεω. Να έχουμε λοιπόν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και την ισορροπία που όλοι επιδιώκουν. Πολύ δουλειά πρέπει να γίνει ακόμη, συμβαστικέ τροπολογίε Θα, τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Κλόντ. Προέδρο, ευχαριστούμε πολύ Ναταλή. Αγαπητοί συνάλφοι, η συζήτηση για τις θεωρήσεις και για τα δικονομικά δικαιώματα είναι μείζωνα θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και για την ε, προσέλευσή τους σήμερα και για την ουσιαστική τους ε, συνεισφορά. Σήμερα, πρωί Πέμπτης, έχουμε πολλά θέματα στη Διάταξη και έχουμε παρατείνει πολλά θέματα. Άρα, το 9 θα το συζητήσουμε την 1η Απριλίου. 1η Απριλίου, το βγάζω δηλαδή το 9 από τη Μεσιαδιάταξη. Διάταξη. Λοιπόν, σημείο 8 τώρα, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Um, Σημείο 8. Παρουσίασε του και προγράμματος εργασίας για το 2015 και παρακολούθηση της αξιολόγησης που δημιουργήθηκε το 2013. Από τον Διευθυντή Μόρτεν Καερούμ και την Πρώτη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάγια Καρίνα Σάξλιν. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε τον Διευθυντή και την Πρώτη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί μας. Θα δώσω στην κυρία το λόγο πρώτα να μας παρουσιάσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού για το 2015 και βέβαια μετά ο Μόρτεν Κάιρουμ θα μας πει ό,τι θέλει να μας πει. Further I'm going to take, uh, take you first and then a Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις εργασίες ε, του Οργανισμού Ανθρωπίνων, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία και υποστήριξή σας. Τώρα που λύγει η θητεία μου ως Προέδρου του ε, Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθυντής μας θα βρει νέες προκλήσεις για το μέλλον του. Ο κύριος Μόρτεν Κέρουμ θα μιλήσει για τα επιτεύγματα του οργανισμού και τις προσπάθειές του να βρει λύσεις στις προκλήσεις που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και που αντιμετωπίζουμε εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα όμως πρώτα να σας μιλήσω για κάποια από τα προγράμματα κλειδιά του οργανισμού. Θα αναφερθώ ε, σε αυτά όπως παρουσιάζονται στο, στην ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και που είναι χωρισμένη σε τρεις τομείς, ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη. Όσον αφορά την ελευθερία στον τομέα της μετανάστευσης, ε, μια εμπληματική δημοσίευση μας φέτος έχει να κάνει με τις σοβαρές μορφές εκμετάλλευσης ε, της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αναφέρονται διάφορα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των θυμάτων και η ελεύθερη κινητικότητα. Πάνω από 600 συνεντεύξεις ε, διεξάγαμε και φαίνεται ότι υπάρχει ένα μοτίβο σύγχρονης σκλαβιάς σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα ε, στην ε, γεωργία, οικοδομές ε, και οικιακές εργασίες και καθαρισμός. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε αρχές Ιουνίου αναφέρεται σε διάφορες οδηγίες όπου χρειάζονται αναθεώρηση ή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, όπως είναι η οδηγία για ε, τα δικαιώματα των θυμάτων. Ε, και θέλουμε να ε, δώσουμε όσο γίνεται περισσότερη ορατότητα στις ανησυχίες που επισημένονται στην έκθεση. Άλλο σημαντικό πρόγραμμα φέτος εξετάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα σε σχέση με την ε, συλλογή και αποθήκευση βιομετρικών δεδομένων ε, για σκοπούς ελέγχου των ε, συνόρων και έκδοσης θεωρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό που βρίσκεται ακόμα στα πρώτα του στάδια τονίζει την συλλογή βιομετρικών δεδομένων από ε, το σύστημα πληροφόρηση σε το σύστημα πληροφόρηση για τις θεωρήσει και την Eurodac. Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος ε, θα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον οργανισμό e και την Frontex και μπορεί να επηρεάσουν και τις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το πακέτο έξυπνων συνόρων, εφιών συνόρων. Είναι ένα θέμα που αφορά τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών και Τις έρευνες αυτές τις κάνουμε κατόπιν ε, αιτήματος ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ μετά το ψηφίσμα του προηγούμενου μήνα για το πρόγραμμα παρακολούθησης ε, του NSA. Η Εθνική φορείς για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Θα προχωρήσω τώρα στον επόμενο θεματικό τομέα στο πρόγραμμα εργασίας μας, την ισότητα. Ρατσισμός, ξενοφοβία, μυσαλλοδοξία και θέματα διακρίσεων ένταξη των Ρωμά και τα δικαιώματα του παιδιού. Οργανισμός ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θέσπισε το πολιετές ε, πρόγραμμα Ρωμά το 2012 κατόπιν ετήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό του προγράμματος, πρόσφατα, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα τοπική συμμετοχή για την ένταξη των Ρωμά που στόχο έχει την ενθάρρυνση των τοπικών κοινωνιών για την ε, εφαρμογή μέτρων ένταξης των Ρώμα σε τοπικό επίπεδο. Θα παρακολου... Μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε μια δραστηριότητα παρακολούθηση των μέτρων του προγράμματος αυτού. Το 2015 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα εξετάσει το θέμα των ατόμων ΛΟΑΔ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, λεσβιών, αμφιλόφιλων, ομοφιλόφιλων κλπ. Και ε, τέτοιοι άνθρωποι ερωτήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις εμπειρίες τους και διαπιστώθηκε ότι η παρενόχληση στα σχολεία και η ομοφοβική βία είναι φαινόμενα εξαπλωμένα. Είχαμε σε με δημόσιες αρχές και με παρόχους υπηρεσιών για να διαπιστώσουμε εάν και κατά πόσο οι πρακτικές και οι πολιτικές σε εθνικό επίπεδο συμβάλλουν στην δημιουργία ε, ίσων ευκαιριών για τους ε, ανθρώπους ΛΟΑΔ. Φέτος θα δημοσιευτούν εκθέσεις και άλλες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτές οι μελέτες μπορούν να σας δώσουν στοιχεία για τις εργασίες σας σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, παράλληλα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 25 ετή για τον εορτασμό της 25 ετίας ε, της ε, Σύμβασης ε, των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Διάφοροι επαγγελματίες του χώρου που συμμετέχουν στις διαδικασίες αλλά και παιδιά ερωτήθηκαν για να εξεταστούν οι εμπειρίες τους σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ποινικέ και άλλες διαδικασίες. Έτσι διαπιστώθηκε σε τι βαθμό οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης εφαρμόζονται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμπεράσματα θα είναι χρήσιμα και για τα κράτη-μέλη σε προετοιμασία της εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων ε, τώρα το φθινόπωρο. Κυρίες και κύριοι, προτού να κλείσω θα ήθελα να... να αναφερθώ στον κανονισμό για τη χρηματοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, για θέματα τρίτου πυλώνα για την αστυνομική συνεργασία σε ποινικά θέματα δεν έχει διασφαλιστεί η ε, το δικαίωμα του οργανισμού να ε, γνωμοδοτεί χωρίς να υπάρχει αίτημα από ένα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ε, εξωτερική αξιολόγηση του οργανισμού, στην οποία θα αναφερθεί ο Μόρτεν πιο αναλυτικά, ε, προβλέπει ότι θα εποφεληθεί ο νομοθέτης από πρωτοβουλίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στον τομέα αυτών. Και μία τελευταία παρατήρηση. Οι εργασία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, εργάζεται πάνω σε θέματα τα οποία μόνο εν μέρη άπτονται των κοινωνικών δικαιωμάτων το διοικητικό μας συμβούλιο θεωρεί ότι για να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πενταετές πρόγραμμά μας ή το πολιετές πλαίσιο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα κοινωνικά δικαιώματα που ε, αφορούν τις κοινωνίες μας. Αυτό θα μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε ε, όσο γίνεται περισσότερο τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός μας θα αυξήσει τη δυνατότητα, τις δυνατότητές του ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα να γίνονται σεβαστά για όλους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον Μόρτεν Κέρουμ, Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Πρωτού δώσουμε το λόγο στους βουλευτές μας για ερωτήσεις. Πριν ακούσουμε τον Μόρτεν, θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέρφους ότι όπως γνωρίζετε και πολλοί από εσά, αυτή θα είναι η τελευταία παρουσίασή του προς την ε, Επιτροπή ΛΥΒΕ. Ήταν διευθυντής από το 2008 που δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εγώ τον ξέρω όσο καιρό είμαι βουλευτής εδώ και θα ήθελα να τον επενέσω ιδιαίτερα διότι είναι πολύ δύσκολο το να διευθύνει κανεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη στιγμή που υπάρχουν και πολύ διστάμενε απόψει σχετικά με το τι είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, έχει ασκήσει τα καθήκοντά του με ε, αίσθημα ευθύνη και θέλω να σα ευχαριστώ για την δουλειά σας σε μια πολύ δύσκολη θέση θα γίνετε διευθυντή σε μεγάλο ερευνητικό οργανισμό στη Σουηδία. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι. Παρακαλώ. Τώρα βέβαια μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε που αποχωρείτε. Παρακαλώ. Thank you very much. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πολύ Κλοντ. Είναι τεράστια ευχαρίστηση για μένα και ήταν τεράστια ευχαρίστηση το ότι μπορούσα και ερχόμουν εδώ πέρα και μιλούσα τόσο συχνά μαζί σα, εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Είχαμε πάντα έναν ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο και πάντα εκτιμούσα πάρα πολύ την ανταλλαγή απόψεων που είχα μαζί σα. Και εύχομαι ότι θα καλωσορίσετε με τον ίδιο τρόπο τον διάδοχό μου και ότι θα εξακολουθείτε να έχετε μαζί του τον ίδιο επικοδομητικό διάλογο που είχαμε μαζί τα πρώτα 7-8 χρόνια του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από προσωπικής πλευράς να πω ότι ήταν ένα καταπληκτικό προνόμιο το ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να στήσω, να δημιουργήσω με τη βοήθεια των συνεργατών μου προφανώς ένα νέο οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να επισφέρουμε μια προστιθέμενη αξία. Τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή ο οργανισμός μας προκειμένου να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και κατ' επέκταση βέβαια τα κράτη-μέλη. Έχουμε καλύψει, θεωρώ, μεγάλη απόσταση. Δημιουργήσαμε έναν οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων που πληρεί πλήρω την ε, εντολή του. Έναν οργανισμό που εξακολουθεί και έχει σημαντική επίπτωση για διάφορα κέρια ζητήματα, όπως φάνηκε άλλωστε και στην εξωτερική αξιολόγηση που μας έγινε το 2013. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αφαιρθώ σε ορισμένα ζητήματα τα οποία επεξεργαστήκαμε και με τα οποία ασχολήθηκε και η εξωτερική αξιολόγηση. Τα τελευταία αυτά χρόνια δημιουργήσαμε μία μοναδική δεξαμενή δεδομένων όσον αφορά κάποια βασικά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήματα για τα οποία οφείλω να πω ότι είχαμε ελάχιστη και καμία γνώση προτού ξεκινήσουμε την εργασία μας. Να αναφερθώ σε ένα για παράδειγμα. Τα εγκλήματα λόγω μίσους, είναι ένα ζήτημα για το, το οποίο γνωρίζαμε ελάχιστα. Το βλέπαμε απλώ να αναφέρεται σε κάποιε έρευνε. Κάναμε λοιπόν κάποιε έρευνε όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών. Συμμετείχαν στην έρευνα αυτή 42.000 γυναίκε. Είχαμε 93.000 συμμετέχοντε στην έρευνα για του ΛΟΑΔ, μια μεγάλη έρευνα για του Ρωμά, όπου συμμετείχαν 80.000 Ρωμά και πολλά νοικοκυριά, μια άλλη έρευνα για τις εθνοτικές μειονότητες και διεξήγαμε επίσης και μια έρευνα όσον αφορά τον αντισημιτισμό, έρευνα η οποία χρησιμοποιήθηκε δυστυχώς πολύ το τελευταίο διάστημα από τα κράτη-μέλη. Υπήρχε πάντως η έρευνα αυτή, διεξήχθη από μας και μας έκανε να καταλάβουμε ποια είναι η εμπειρία της εβραϊκής κοινότητας σε διάφορες χώρες, σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι έρευνες λοιπόν μας διαφωτίζουν για διάφορα ζητήματα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων και χάρη στις έρευνες αυτές θεωρώ ότι και εσείς καταφέρατε να στοχεύσετε καλύτερα την νομοθεσία την οποία επεξεργάζεται εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από όλα αυτά βέβαια, προχωρήσαμε και σε μια σειρά νομικών αναλύσεων και μελετών ε, εκδώσαμε διάφορα εγχειρίδια τα οποία ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή. Ε, κάποια έχουν εξαντληθεί 150.000 περίπου αντίτυπα έχουν ε, διανεμηθεί για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διακριτική μεταχείριση, για τα δικαιώματα των προσφύγων και των ασύλων, για τα δικαιώματα των παιδιών, οδική και εγχειρίδια, τα οποία εκπονήσαμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και οφείλω να πω ότι είχαμε μια πολύ θετική συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και είμαι ιδιαίτερα περήφανος όταν σας λέω ότι η έκθεσή μας η οποία διανεμήθη, μάλλον η έκθεσή μας, η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ήταν η πιο δημοφιλή, από τις πιο δημοφιλείς εκθέσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχουν 300 βασικοί ενδιαφερόμενοι στον Οργανισμό Θεμελιών Δικαιωμάτων. Αναφέρομαι βέβαια σε διάφορου οργανισμού εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών, αλλά και στέλνει τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαφώς υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την ε, δράση μας και όπως μόλις τώρα υπόθηκε από τη συνάδελφό μου, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα νομικών γνωμοδοτήσεων, δηλαδή να μπορούμε κι εμείς να συμβάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο στη δική σας νομοθετική διαδικασία, να μπορούμε στοχευμένα να επεμβαίνουμε. Δυστυχώς είμαστε πολύ περιορισμένοι όσον αφορά το δικαίωμα νομικής γνωμοδότησης. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες βέβαια που μα δόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίω όταν έρχεστε έρχεστε σε εμά και μας ζητάτε συγκεκριμένη περιστατωμένη γνωμοδότηση για συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία επεξεργάζεστε, αλλά θα θέλαμε από την άλλη να μπορούσαμε και εμείς με δική μας πρωτοβουλία να υποβάλουμε γνωμοδοτήσεις για διάφορα ζητήματα χωρίς απαραίτητα να μας το ζητά ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρόμαστε πάντως πολύ που βλέπουμε ότι όλες οι μελέτες και έρευνες που έχουμε εκπονήσει χρησιμοποιούνται τελικά στην πράξη κατά την εκπόνηση κοινοτική νομοθεσίας. Δεύτερον, ένα ακόμα ζήτημα στο οποίο θεωρώ ότι μπορεί να επέλθει μια κάποια βελτίωση είναι το ζήτημα των γυναικών. Ξέρετε ότι ε, ασχοληθήκαμε με το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών του οργανισμού μας και τα τελευταία χρόνια ως ε, οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταφέραμε να συνεργαστούμε πιο έντονα με τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ζητήσαμε σε θελούσια βάση να διορίζουν στο κοινοβούλιο τους ένα σημείο επαφής, ένα focal point, το οποίο θα αποτελούσε σημείο σύνδεσης ανάμεσα στον δικό μας τον οργανισμό και τα εθνικά κοινοβούλια. Δείξαν θετική στάση όλα σχεδόν τα κοινοβούλια και ήρθαν στη Βιέννη την προηγούμενη εβδομάδα όπου είχαμε μια κοινή συνεδρίαση ανταλλαγής απόψεων τόσο για το πώς θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε αυτή τη συνεργασία αλλά συζητήσαμε και για την συνεργασία, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα για τα οποία γνωμοδοτεί η ΦΡΑ, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πιέζει ο χρόνος να αναφερθώ σύντομα σε δύο-τρία ζητήματα, τα οποία θεωρώ ότι αξίζει να θίξουμε. Πρώτον, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο όσον αφορά το ζήτημα της κατανόησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως οριζόντιο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, πολύ συχνά, κάθε φορά που με ρωτάνε για ποιο λόγο δεν ήσασταν προσκεκλημένοι στη μία ή την άλλη συνεδρίαση. Πολύ συχνά η απάντηση είναι ότι μα, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούσαν ζήτημα στη μερίσια διάταξη, μολονότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση μπορεί οι βουλευτές, οι άλλοι συμμετέχοντε να συζητούσαν ζητήματα που άπτονται του ασύλου, των προσφύγων, των Ρωμά κτλ. Ουσιαστικά ζητήματα τα οποία έχουν μια πολύ σημαντική συνιστόσα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε λοιπόν να μην απομονώνεται το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην, να θεωρείται παράτερο ξεχωριστό ζήτημα, αλλά συνειδητοποιήσουμε ότι όντω αποτελεί οριζόντιο ζήτημα πάρα πολλών θεμάτων τα οποία θίγουμε. Επίσης, η Ιταλική Προεδρία επέμεινε πάρα πολύ στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας. Πάντως όχι μόνο στα νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια αλλά και στα υπόλοιπα νομοθετήματα θα πρέπει πάντα να τονίζεται η πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως επανερχόμενο στο ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να σας πω ότι η συνιστόσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα θα υπάρχει. Ξέρετε ότι πάντα μιλάμε για ήπιο δίκαιο ή πιο σκληρό δίκαιο soft hard Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε περισσότερο για smart προσέγγιση, για ευφυή προσέγγιση όσον αφορά την συνιστόσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίω για την εσωτερική ασφάλεια. Πώ θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρί αποκλεισμού, μια κοινωνία η οποία θα είναι πιο συνεκτική. Και ξέρετε ότι στα πλαίσια του οργανισμού μα έχουμε πολλέ μελέτε που όντως φωτίζουν πολλές προκλήσεις που δεν έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει και πάρα πολλά ζητήματα όπως το ethnic profiling, το κατάρτιση προφίλ με βάση την εθνοτική προέλευση, ζητήματα τα οποία δεν συμβάλλουν τελικά στη δημιουργία συνεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλήσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Επανερχόμενος τώρα στο τρίτο ζήτημα Πρέπει να σας πω ότι ταξίδεψα παντού στην Ευρώπη τα τελευταία 7 χρόνια και βλέπω ότι υπάρχει μία οργή που όλο και μεγαλώνει. Μία οργή που προέρχεται από τους πολίτες. Η οικονομική κατάσταση, τα μέτρα λιτότητας έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη απόγνωση στους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή ένα πλαίσιο προάσπισης των κοινωνικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πραγματικά λυπηρό που ο οργανισμός μας δεν κατάφερε να έχει συγκεκριμένη εντολή όσον αφορά το ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ασχολούμεθα με το ζήτημα αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να το ενισχύσουμε λίγο περισσότερο και να μπορούμε να είμαστε περισσότερο αρμόδιοι για το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά το άσυλο, χρειαζόμαστε προφανώς μια πιο υψηλόβαθμη αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά το ζήτημα του ασύλου. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω τη σημασία της συμβολής των θεσμικών οργάνων στη δράση την οποία εμείς αναλαμβάνουμε, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συνειδητοποιήσουμε τη συλλογική μας ευθύνη. Συλλογική πρέπει να, πρέπει να είναι η δράση μας, συλλογικά θα πρέπει να κυνηγούμε τους ίδιους στόχους, συλλογικά θα πρέπει να καταφέρουμε να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δημιουργήσουμε ένα υψηλό βαθμό επίπεδο προάσπισης τους. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε μια συνοχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνοχή πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επ' αυτού πολλά πράγματα ακόμα μπορούν να γίνουν για να δημιουργηθεί περισσότερη συνεργασία, συμπληρωματικότητα ανάμεσα στου διάφορου εμπλεκόμενου και στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σημειώσει πάντω σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια Πάντως ελπίζω και με τον νέο διευθυντή που θα με διαδεχθεί να έχετε την ίδια επικοδομητική συνεργασία που, καταφέραμε, που καταφέρατε να έχετε μαζί μου. Και προφανώς βέβαια απομένουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Σας εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια για το μέλλον και ελπίζω ότι θα καταφέρω να σας δω τους μεν και τους δε και στο μέλλον, ακόμα και αν δεν συνεχίζω να είμαι διευθυντής βέβαια αυτού του οργανισμού. Ναι, έχει περάσει πολύ καιρό. Και είναι πολύ δύσκολο να χειριστεί κανεί και όλε τι προσδοκίε από το πρόσωπό σα. Σα ευχαριστούμε πολύ για τι υπηρεσίε σα. Στο όνομα όλων των μελών της ΛΥΠΕ που έχουν συνεργαστεί μαζί σας, ε, μερικοί είναι απόντες, άλλοι παρόντες. Έχουμε λοιπόν αρκετές ερωτήσεις, 20 λεπτά στα οποία μπορούμε να σας θέσουμε τις ερωτήσεις αυτές. Και είναι πολύ δύσκολο το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να χειριστούμε τα θέματα αυτά. Ε, την αντιτρομοκρατία, για παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ε, θα θέσω εγώ τις ερωτήσεις αυτές. Ε, να ρωτήσω τα μέλη της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι όλοι κουράστηκαν. Είχαμε ήδη δύο πολύ σημαντικές συζητήσεις σήμερα το πρωί. Συνάδελφοι, ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει, παρακαλώ. Silly of course we have very ναι, είμαι ανόητος αφού έχουμε εδώ ήδη μια, ένα κατάλογο με εκατοντάδες ονόματα. Συγγνώμη. Καινούριο είμαι. Κυρία Ντάτη, θέλετε το λόγο παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, καταρχά σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σα, καθώ επίση και για το σημαντικότατο έργο το οποίο επιτελέσατε στα πλαίσια του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στα φιλόδοξα σχέδια, τα φιλόδοξα προγράμματα τα οποία προωθήσετε στα πλαίσια του οργανισμού σας. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, η προστασία των θεμελιωδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας αφορά όλους και όλες τις πολιτικές ομάδες. Μπορούμε να έχουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικούς τρόπους προάσπισής τους, πάντως τα θεμελιώδη, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Αποτελεί κοινό μέλημά μας. Είδα το πρόγραμμα εργασία για το 2015 και θα ήθελα να επιμείνω σε δύο σημεία και θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μα είπατε ότι γίνεται ένα σημαντικότατο ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να παρακάμψουμε, ιδίω στα πλαίσια τη παρακολούθηση μεγάλη κλίμακα και επίση το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπω είπατε και εσεί, γίνεται πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω σε, περί... περίοδο οικονομική κρίση και όταν οξύνονται τελικά οι ανισότητε μεταξύ των χωρών και των πολιτών. Θεμελιώδη δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες είναι δύο έννοιες που συνάδουν. Αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε εμείς να αναλύσουμε κάθε φορά που συζητούσαμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η έκθεση την οποία υποβάλλεται για το 2015 είναι πάρα πολύ θετική και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό που βλέπουμε ότι μέσω της δική σας της δράσης καταφέραμε να έχουμε τα απαραίτητα εχέγγυα για την προστασία της προσωπικής ιδιωτικής ζωής χωρίς όμως να θυσιάζουμε και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς να βάλουμε κατά του πολύ αποτελεσματικού και αναγκαστικού έργου που επιτελούν οι υπηρεσίες μυστικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς όμως ποτέ να οδηγούνται σε κατάχρηση αυτή τη εξουσία του. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάτι που αναφέρατε κι εσείς, εκπόνηση εγχειριδίου όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγχειρίδιο που αναφέρεται στην ένωμη τάξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και στην υφιστάμενη νομολογία που επιτρέπει στους πολίτες να καταλάβουν ποια είναι τα δικαιώματά του πρόσβαση στη δικαιοσύνη η κυρία Μόνικα Χολμάιρα αναφέρθηκε επίση αυτό πριν από λίγο. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθίσταται περίπλοκη για πάρα πολλού πολίτες τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Κύριε Διευθυντά, οι δράσει σας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία, την πιο αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματο. Πολλέ φορέ μα είπατε ότι στα πλαίσια μια δίκη τα θεμελιώδη δικαιώματα καταπατώνται. Εμεί θεωρούμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα προφανώ θα πρέπει να προασπίζονται πλήρω στα πλαίσια οποιασδήποτε δικαστική διαδικασία που αφορά οποιονδήποτε πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Λόπεθ Αγιλάρ, που ήταν και πρόεδρος Επιτροπής μας ε, το μεγαλύτερο μέρο της θητείας σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κλόντ, ευχαριστώ Μόρτεν, χαίρομαι που σε βλέπω και που σε είχαμε σε αυτή τη θέση. Είναι προφανές ότι έχουμε υπερβεί ε, το χρόνο μας, αλλά και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έκανε τη διαφορά και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλω να σε ευχαριστήσω και για τις ετήσιες εκθέσεις που μας διαβίβαζες και γιατί ήσουν πάντα ε, μέσα στα χρονοδιαγράμματα και για τα πιο ε, επίγοντα ζητήματα. Η υποβάθμιση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας στην Ήπειρό μας που πρέπει ε, η πυρός μας να είναι η οικογένεια της δημοκρατίας, ο πατέρας και η μητέρα της δημοκρατίας. είπε όμως ε, ότι είχαμε μια τεράστια, τρομερή διαχείριση της κρίσης, ε, υπό αρνητική έννοια πάντα. Και αυτό οδήγησε στο να ξαναβγούν στην επιφάνεια πικρίες κυρίως γιατί αυξήθηκε η οικονομική ανισότητα, όλοι να ζητούν από τράγους. Και έχουμε δει λοιπόν ομοφιλοφοβία, ξενοφοβία, εθνικισμούς, αντισημιτισμό κατά των ε, τσιγκάνων και των Ρωμά. Ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ε, ρίχνοντας το φως των προβολέων στις προκαταλήψεις τη διακριτική μεταχείριση. Και σε όλες τις πολύ γνωστές μορφές, σε όλους αυτούς τους δαίμονες που τόση αματοχυσία και τόση καταστροφή έχουν φέρει. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που συνθέτουν το πάζλ αυτού, αυτό και του αντισημιτισμού. Παραλαμβάνω, επανέρχονται παλιές προκατάληψεις κατά των Εβραίων που τους παρουσιάζουν ως συνομότες. Γενικώ υπάρχουν πολλές θεωρίες νομοσιολογίας και πολλές φορές παίρνουν το ρόλο του αποδιακομπέου τράβου σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ ανησυχητικό που θα πρέπει να μας ανησυχεί ως φαινόμενο. Φυσικά πάλι εθνικισμός, αλλά έχουμε και τον τζιχαντισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση των τζιχαντιστών Ισλαμιστών που αναζητούν τους θήτες στο πρόσωπο των Εβραίων. Ήταν κάτι που μπορεί να ήταν κάτι που βλέπαμε πριν από κάποιες δεκαετίες, το να μπει σε ένα εβραϊκό εστιατόριο σε μια συναγωγή και να σκοτώνεις αθώους ανθρώπους για να κάνεις μία δήλωση, να πεις κάτι. Ε, αυτό το ξαναβλέπουμε τώρα. Φυσικά το μίσος και το έγκλημα και ιδίως online και η παρότρινση σε μίσος και στην ε, τέλεση εξώπινων Αυτό το βλέπουμε online πλέον, στο διαδίκτυο. Cyber hatred κυβερνομίσος μπορούμε να το αποκαλέσουμε. Είναι εικονικό φαινόμενο, όχι όμως και το μίσος. Το μίσος είναι πραγματικό. Απλά κρύβονται αυτοί οι δίληπες από την ανωνυμία. Πίσω από ψεύτικα πρόσωπα, συγκαλύπτοντας, κρύβοντας την ταυτότητα, την πραγματική. Αλλά παρόλα αυτά αυτός ο ποταμός μίσους που χύνεται στο διαδίκτυο είναι πραγματικός. Αυτός ο τζιχαντισμός, αυτή η ριζοσπαστικοποίηση βλέπουμε ότι κερδίζει όλο και πιο πολλούς νέους που είναι απογοητευμένοι, που είναι αγανακτισμένοι, περιθωριοποιημένοι. Περνάνε όλη τους τη ζωή στο ίντερνετ και ρίχνουν μίσος και επιτίθενται στους πλησίον τους ζητούν εκδίκηση κατά των θητών και αυτών που αδικούν τους συμπολίτες τους. Μόρτεν, σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Um, next is Judith Judith. είναι επόμενη. And my colleague uh, Ulrike Lunacek just whispers, and please say... Μου ψιθυρίζει η Ουλρίκε να πω και εκ μέρους της ευχαριστώ. Αυτό να ξεκινήσω λοιπόν. Σας ευχαριστούμε και οι δύο και τους δύο που βάλατε τα θεμελιώδη δικαιώματα στην κορυφή της ατζέντα. Είναι σίγουρα δύσκολο ως πολιτικοί να αποστρέψουμε το βλέμμα σε από αυτά τα θέματα. Άκουσα τις προτάσεις σας για το επόμενο έτος, μάλλον για το τρέχον, το 2015. Πρέπει να πω ότι ε, με συνεπήραν αυτά που είπατε και έχω να διαβάσω πολλά. Προστασία δεδομένων, μετανάστευση. Πολύ ενδιαφέρον μου φαίνεται. Επειδή δεν θέλω να με μακρηγορήσω, ε, θέλω να τονίσω ένα στοιχείο από αυτόν τον κατάλογο που μας ε, αναφέρατε για το 2015. Και μιλώ για την οδηγία περί δικαιωμάτων των θυμάτων και την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και το άρθρο 1 που λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία δικαιωτική μεταχείριση. Δηλαδή, αν κάποιος διαμένει στη χώρα, ε, ε, πρέπει να έχει σεβαστά τα δικαιώματά του, ανεξαρτήτως, λέει, του τρόπου διαμονής. Δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Στη δική μου χώρα, την Ολλανδία, δεν υπάρχει η διάταξη αυτή. Αλλά πρέπει να υπάρχει. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν, όταν εξετάσετε αυτό το ε, θέμα, να μας πείτε ποιες χώρες δίνουν δικαιώματα σε αυτούς τους μη νομίμως διαμένοντες όταν είναι θύματα, σε μια, ε, θύματα μιας αξιόπινης πράξης. Ο Πρόεδρος. Δεν είναι απλά εκθέσεις που ε, μετά μπαίνουν σε ένα ντουλάπι, σκονίζονται σε ένα ράφι, αλλά μιλάμε για πραγματικές ε, περιπτώσεις ε, υλοποίησης. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αλόν Θα σας μιλήσω αφού σας συγχαρώ και για τα καθήκοντα. Για την τρομοκρατία που μίλησε και ο Κλόντ Μωρέ πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη πρέπει με προστατευτικά μέτρα να προστατέψουν του πολίτε και ε, την ασφαλειά του και τι θεμελιώδει του ελευθερίε. Πρέπει να βρεθεί αυτή η σημαντική ισορροπία. Και εμεί στο Κοινοβούλιο υιοθετούμε μια συνολική προσέγγιση, συμπληρωματικά δηλαδή, πρόληψη ρίζοσπαστικοποίηση και μέτρα ασφάλεια. Βέβαια πρέπει και τα θεμελιώδη δικαιώματα να συμπεριληφθούν και στην ε, χάραξη και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Πάντα είναι πολύτιμη συμβολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, μας βοηθά στο νομοθετικό έργο. Δύο ερωτήματα. Μπορέστε ήδη να, έχετε, να γνωμοδοτήσετε, τέλο πάντων να εγγύψετε στο νέο σχέδιο έκθεση του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό PNR που υποβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω μήπως είναι λίγο πρόωρο. Και το δεύτερο ερώτημα πώς με βάση τον οργανισμό μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκπόνηση μέτρων για την καταπολέμηση του λόγου μίσους, ε, ιδίως στο διαδίκτυο. Αυτό θα ρωτήσω και εγώ. Δράτω μου λοιπόν της ευκαιρίας να θέσω να πάρω μια ερώτημα. αν έπρεπε να δώσετε κάποια συμβουλή στον διάδοχό σας, ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή σε σχέση με το νέο πλαίσιο, στο πλαίσιο της ασφάλειας. Σίγουρα είναι άκρος πολυπλοκή κατάσταση. Δεσμευόμαστε νομοθετικά να εστιάσουμε στα συστήματα του PNR και το καθεξής, γιατί αυτή είναι νομοθεσία. Δυστυχώς όμως, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, πάντα ε, αυτό που προέχει είναι οι βέλτιστες πρακτικές και όχι τόσο η νομοθεσία. Δύσκολο το πλαίσιο λοιπόν. Άρα για τον οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τι συμβουλή θα δίνατε, ποιος είναι ο ρόλος του οργανισμού, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Το νέο διοικητικό συμβούλιο, πώς θα του λέγατε να αντιμετωπίσει το πολύ λεπτό αυτό ζήτημα, δεν είναι εύκολο το ερώτημα. Θα ήθελα να ακούσω όμως την προσέγγισή σας και τι θα ζητήσατε και από τα, κράτη, ε, από τα, συγγνώμη, από τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σίγουρα πάντα στα πρωτοσέλιδα μπαίνουν ε, τα νομοθετήματα για προφανείς λόγους, αλλά πώς θα βρούμε αυτή την ισορροπία, πώς θα την πετύχουμε. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Is, um, Στον κατάλογο τώρα, τελευταία ομιλήτρια, η Σόφιν Τβέλτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομη. Πρώτα απ' όλα, Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κύρουμ για την πολύ καλή συνεργασία που διατήρησε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσα χρόνια ήταν επικεφαλής του οργανισμού. Το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Η ομάδα μου θα ήθελα να υπάρχουν πιο πολύ δεσμευτικά μέτρα για την επιβολή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους και της δημοκρατίας ένα σύμφωνο δημοκρατικής διακυβέρνησης προτείνουμε. Διότι γνωρίζουμε ότι δεν σέβονται όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενίοτε μάλιστα βλέπουμε σοβαρές συστηματικές παραβιάσεις. Και ποτέ δεν ενεργοποιείται το άρθρο 7. Δυστυχώς, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατηγορηματικά απέρριψε την πρόταση για οποιοδήποτε νέο μέσο. Πιστεύει ότι ο διάλογος και η σιωπηρή διπλωματία είναι η λύση. Εσείς θα ήσασταν υπέρ δεσμευτικών μέσων και εργαλείων πιο πολύ με βάση τη δική σας εμπειρία ή και εσείς πιστεύετε ότι ο διάλογος και η διπλωματία αρκούν. Έρχομαι τώρα σε ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα, αν κατάλαβα καλά. Ε, είναι ο τελευταίος μήνας σε αυτή το αξίωμα. Από 1η Απριλίου θα ασχοληθείτε με πιο ευχάριστα πράγματα, ελπίζω τουλάχιστον. Ερώτημα λοιπόν, ε, σας το έκανε και ίσως και ο Πρόεδρος. Η διαδικασία ορισμού του διαδόχου ολοκληρώθηκε, πόρο απέχει από την κατάλαβα. Είστε αισιόδοξο ότι θα υπάρχει κάποιος στη θέση σας εγκαίρος. Τέλος, τι συμβουλή θα δίνετε εσείς στο διάδοχό σας για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του οργανισμού. Δεν νομίζω ότι είναι εντός θέματος ε, η πρώτη τελευταία ερώτηση ε, την ε, διαγράφω. Μα τέθηκε, λέει η κυρία Εντβέλτ, και δεν πρέπει η Επιτροπή μας να γνωρίζει αφού θα γίνει ακρόαση με τους υποψηφίου εδώ λοιπόν, κύριε Κύρουμ, ε, κάντε ό,τι θέλετε, ε, δώστε τα όλα, κάντε όπως θέλετε όμως εσείς γιατί η τελευταία σας εμφάνιση εδώ. Αποφασίστε οι δυο σας ε, τι θα κάνετε, πώς θα μιλήσετε, τι θα απαντήσετε. Νομίζω ότι και τα διδάγματα που έχετε αντλήσει και το τι συμβουλές θα δίνατε στο διάδοχό σας είναι από τα βασικά ερωτήματα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας και τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις σας, ιδιαίτερα προς τον Μόρτεν. Είμαι βέβαιη ότι και αυτή η συζήτηση θα βελτιώσει τη, τη δουλειά μας. Ε, νομίζω θα αφήσω τον Μόρτεν να απαντήσει. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καταρχάς να σας ευχαριστήσω για όλα τα ευγενικά σας λόγια. Όπως είπα στην αρχή και από πλευράς μου ήταν χαρά να συνεργαστώ με πολλούς από σούς ε, κατά τη διάρκεια μια μισής ε, θητείας. Όσον αφορά τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και να περάσω μετά στις συμβουλές που θα έδινα στο διαδοχό μου. Η κυρία Ντατή αναφέρθηκε στο θέμα της προστασίας δεδομένων και στο θέμα ασφαλείας και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέλουμε και εμείς να τονίσουμε ότι πρόκειται για δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος μετά την 11η ε, Σεπτεμβρίου ε, τέθηκε η συζήτηση ότι είτε θα έχουμε θεμελιώδη δικαιώματα είτε θα έχουμε ασφάλεια, αλλά θεωρούμε ότι ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να είναι σημαντικό κομμάτι οποιασδήποτε πολιτικής ασφαλείας. Πιστεύουμε ότι τα θέματα αυτά είναι άμεσα συνδεμένα μεταξύ τους. Προκλήσεις τις οποίες θα αναλύσει ο οργανισμός μας εντός της άνοιξης και του καλοκαιριού. Κάτι που έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο είναι οι μηχανισμοί προσφυγής. Νομίζω ότι όταν δίδονται τόσες αρμοδιότητες στις υπηρεσίες ασφαλείας θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και μηχανισμοί προσφυγής διότι για παράδειγμα με τις νέες τεχνολογίες έχουν τεράστιες δυνατότητες, γι' αυτό χρειάζεται αυτές οι δομές να ενσωματωθούν στο σύστημα. Σε πολλά κράτη-μέλη είναι πολύ ελλειπείς οι μηχανισμοί προσφυγής, εάν υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν αυξανόμενη ανισορροπία την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε και να μην γελιόμαστε. Προσπαθούμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα με καινούριε μεγάλε βάσει δεδομένων. Πόσο βελτιώνουν ε, τη συνολική ασφάλεια. Ε, εν αυτό θα το εξετάσουν η αστυνομία και άλλοι εμπειρογνώμονε. Αλλά η δική μα ανησυχία από πλευρά των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ότι γίνονται πολλά λάθη. Ο καθένας από εμά λοιπόν μπορεί να καταλήξει σε αυτά τα αρχεία, κάτι που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή μας, την επαγγελματική, τις μεταφορές ή άλλες πτυχές. Τι μηχανισμοί προσφυγής υπάρχουν λοιπόν. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί και μπορούμε να επιμείνουμε να διορθωθούν. Υπάρχουν λοιπόν εδώ διάφορα θέματα τα οποία συνδέονται με τα θέματα αυτά. Στον κύριο Αγγιλάρ, να πω ευχαριστώ για, τις, ε, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ε, όσον αφορά τον αντισημιτισμό στον οποίο αναφερθήκατε, ένα από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που είδαμε όταν λάβαμε τα σχετικά δεδομένα ήταν ε, το υψηλό επίπεδο φόβου που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει στις αντίσεις της εβραϊκής κοινότητας σε τρεις χώρες το 40 με 50% όσων απάντησαν είπαν ότι είχαν σκεφτεί σοβαρά να αποχωρήσουν από τη χώρα λόγω της κατάστασης ασφαλείας στη χώρα. Το 2013 μάλιστα πριν τα γεγονότα στην Τουλούζη, στο Παρίσι, στην Κοπεχάγη και στις Βρυξέλλες. Θέλουμε λοιπόν να επαναλάβουμε του χρόνου την μελέτη αυτή το 2016 και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν. Ο φόβος των ανθρώπων. Να μην ξεχνάμε όμως ότι και στην Ισλαμική κοινότητα υπάρχει επίπεδο φόβου το οποίο διαπιστώσαμε πιο επιφανειακά θα έλεγα ε, διότι δεν είχαμε ακόμα εκπονήσει τέτοιες μελέτες. Εκπονήσαμε όμως μία μελέτη γρήγορα ε, μετά τα γεγονότα στο Παρίσι. Αυτή η μελέτη όμως θα γίνει το 2016 που θα επαναλάβουμε την πρώτη μας μελέτη για τις μειονότητες. Έτσι θα συγκεντρώσουμε πολλά δεδομένα και για ε, τον μουσουλμανικό πληθυσμό στην Ευρώπη και τους φόβους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το επιγραμμικό ε, έγκλημα μίσους, κάτι που ανέφερε ο κύριος Αγγιλάρ, ε, που αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. είναι τεράστιο πρόβλημα όπως τονίσατε και οι δυο σας. Δεν έχουμε λύσεις στο θέμα αυτό. Μόλις τώρα ξεκινήσαμε τις εργασίες. Αυτή τη στιγμή ο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν έχει πολλά να προσφέρει. Βρίσκεται όμω το θέμα στο θεματολόγιο μου και προσλέπω στη συνεργασία μαζί σα, διότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Το διαπιστώσαμε αυτό στην μελέτη μας για τον αντισημιτισμό, για τα άτομα ΛΟΑΔ και για τη βία εις βάρος γυναικών. Διαπιστώσαμε δηλαδή ότι το, μίσος, το κυβερνομίσος ε, είναι πολύ σοβαρός παράγοντας και δημιουργεί πολύ έντονο φόβο. Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, Και να μην ξεχνάμε ότι θέλουμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία λόγου και τις δυνατότητες που δίνει το διαδίκτυο από τη μία και από την άλλη την απαγόρευση να παρακινεί κανείς άλλους σε μίσος και έγκλημα. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρούμε την ισορροπία και να έχουμε πιο αποτελεσματική αστυνόμευση. Μας εξέπληξε το μίσος κατά γυναικών τα κοινωνικά μέσα και το πόσο αργά αντέδρασαν οι αρχές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο επίπεδο μίσους που διαπιστώνεται εκεί. Μπορείτε λοιπόν να βασιστείτε στον οργανισμό μας και μάλιστα είναι μία από τις συμβουλές που θα έδινα στον νέο διευθυντή. Οι άνθρωποι χωρίς έγγραφα και τα θύματα. Η οδηγία για τα θύματα. Η οδηγία αυτή είναι ένα από τα σημαντικότερα νομοθετήματα που αποκτήσαμε τα τελευταία χρόνια μπορεί να γίνει πολύ σημαντικό εργαλείο για την παροχή υποστήριξη στα θύματα. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Πολύ λίγα έχουν γίνει όμως. Συνήθως ε, απλά δίδονται πιο αυστηρές ποινέ στου δράστε, αλλά αυτό δεν προστατεύει και τα θύματα. Ο οργανισμός μας λοιπόν έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα των μεταναστών χωρίς έγγραφα. Σας ευχαριστώ που επιστήσατε την προσοχή μου στο θέμα αυτό. Θα εξετάσουμε το θέμα, θα το εξετάσει φυσικά και η Κομισιόν όταν εξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας αυτής ε, και η Κομισιόν που είναι παρούσα. Πιστεύω ότι άκουσε προσεκτικά τα όσα είπατε. Σύμβουλες προς τον διαδοχό μου σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια. Θα ήθελα να του πω να συνεχίσει να συμμετέχει στις συζητήσεις για την εσωτερική ασφάλεια. Δηλαδή και εδώ σε, τούτο τον χώρο, αλλά και στις ε, ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, να συμμετέχει στις, και να επιμείνει να καλούμαστε στα άτυπα Συμβούλια Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Ενώ είχα πολύ καλές σχέσεις με την Ιταλική Προεδρία, απογοητεύτηκα που τον Γενάρη δεν προσκληθήκαμε στο άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών όταν ήταν το συγκεκριμένο θέμα ε, στην ημερήσια διάταξη. Πιστεύω ότι αυτό ήταν λάθος μήνυμα. Όσον αφορά τον ρόλο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις μελέτες που εκπονούμε. Τις αξίες που διακυβεύονται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι θέματα που εξετάζουμε και αυτό είναι κάτι που επιδεινώνει την ε, θέση των μειονοτήτων στην Ευρώπη. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να θέτουμε κέρια ερωτήματα. Η συμβουλή μου λοιπόν θα ήταν στενή συνεργασία με σας, να σας δίνουμε αυτά που χρειάζεται να γνωρίζετε, να εξετάζουμε πού χρειάζεται να γνωρίζετε περισσότερα. Να συμμετέχει ο οργανισμός μας ε, στην νομοθετική δουλειά και να γνωμοδοτούμε, όπως για παράδειγμα στο θέμα των δεδομένων των επιβατών, PNR. Δεν μα ζητήθηκε ακόμα να γνωμοδοτήσουμε στο θέμα αυτό, έτσι δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε επίσημα, αλλά όπω και εσεί ανησυχούμε και εμεί για το θέμα αυτό. Αν θα θέλατε να στείλετε επίσημο αίτημα προ τον οργανισμό μα, είμαι βέβαιο ότι πολύ ευχαρίστω θα γνωμοδοτήσουμε όπω κάναμε το 2008 και το 2011, γιατί λοιπόν όχι και τώρα το 2015. Τέλος, ξέρω, ξέρω, μας πιέζει ο χρόνος. Ξέρω ότι αγχώνεστε. Η Σοφή Νετφέλτ ε, ε, αναφέρθηκε στο θέμα ενός θεσμευτικού οργανισμού. Θα πρέπει να ασχοληθούν πολύ περισσότερο ε, με το κράτος δικαίου. Τι να κάνουμε, χρειαζόμαστε καινούργια εργαλεία. Όχι, εγώ θα έλεγα να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα εργαλεία που έχουμε συμπεριλαμβανομένου του οργανισμού. Θα θέλαμε δηλαδή ενισχυμένο ρόλο του οργανισμού. Δεν θα ήθελα να δημιουργήσουμε νέους φορείς, ε, νέους θεσμούς, αλλά να εκμεταλλευτούμε ε, στο έπακρον αυτά που ήδη υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου είναι δραματική και θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα στον τομέα αυτών. Είναι κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί όλους μας και πρέπει να είναι κάτι το οποίο ανησυχεί όλους μας. Θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλάω, όπως γνωρίζετε, αλλά μάλλον θα πρέπει να κλείσω εδώ. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία μαζί σας και στην ε, νέα μου ιδιότητα. Um, να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά, Μόρτεν. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα σου θέση. και για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να περάσουμε στο επόμενο και τελευταίο σημείο τη ημερησία διάταξη. Να ζητήσω συγγνώμη από τον εισηγητή κύριο Λέραρ που το έχουμε στριμώξει αυτό το θέμα. Είναι ενδιαφέρον όμω το ζήτημα της Λειτουργικότητας για τι ευρωπαϊκές Δημοσιαστικές επιχειρήσει επιχειρήσεις και Πολίτε. Σχέδιο γνωμοδότηση συντάξει ο κύριο Γερούν Λέναρ. Αμέσω σα δώσω το λόγο και λυπούμε πολύ που είναι τόσο σύντομο το διάστημα που έχετε στη διάθεσή σας. Θα είμαι πολύ σύντομος και θα τα πω και στα Ολλανδικά. Το ζήτημα αυτό το έχουμε ήδη συζητήσει. Είχαμε πει ότι από τη μια έχουμε τις κυβερνήσεις, από την άλλη τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ότι η σχέση αυτή όλο και ψηφιοποιείται, όλο και εξυγχρονίζεται και προφανώς υπάρχουν κάποια προνόμια και ωφέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αλλά από την άλλη έχουμε μπροστά μας πολλά διαφορετικά συστήματα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα διαλειτουργικά. Πρέπει λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν ακόμα και διασυνοριακά τα συστήματα αυτά, χωρίς να αντιμετωπίζουν εμπόδια και προβλήματα. Δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί ο ευκταίος βαθμός διαλειτουργικότητος, και κυρίως δεν έχει επιτευχθεί η απαραίτητη προστασία των δεδομένων. Η προστασία λοιπόν των δεδομένων θα πρέπει να διασφαλίζεται στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας αυτής. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να καλύπτεται στη δική μας τη γνωμοδότηση κυρίως αυτό το ζήτημα, καθότι αποτελεί ουσιαστικά καθήλυν δική μας αρμοδιότητα η προστασία των δεδομένων. Γίνεται λοιπόν μια αναφορά στο κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Στην τελογική σκέψη της έκθεσης αναφερόμαστε επίσης στην προστασία αυτών των δεδομένων, στις βασικές αρχές που τη διέπουν. Λέμε ότι έχουμε συγκεκριμένη σωρευμένη εμπειρία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, η οποία θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη και λέμε επίση ότι θα πρέπει να διασφαλίζουμε την τήρηση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων. Μια σημαντική παράληψη βέβαια μέχρι στιγμή ήταν ένα άρθρο. Υπάρχει ένα άρθρο στο ίδιο το διατακτικό τη πρόταση, όπου πραγματικά να γίνεται σαφή αναφορά στην προάσπιση τη αρχή τη προστασία των δεδομένων. Γι' αυτό το λόγο εμεί συντάξαμε ένα νέο άρθρο, το οποίο και λέμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κύριο τμήμα τη πρόταση. Βασιζόμαστε επίσης στο, στην πρώτη μορφή του προγράμματος, το ISA 1. Το 2016 θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο πρόγραμμα, το ISA 2, πρόγραμμα λύσεων διαλειτουργικότητας για τις δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρώπης. Προσβλέπω επίσης και στις αντιδράσεις τώρα των συναδέλφων και σε μία επικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστούμε κύριε Λέναρτς. Ήσταν όπως πάντα ιδιαίτερα γρήγορος και σύντομος στην παρέμβασή σας. Ο πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς. Έχουμε μόνο μία σκιώδη εισηγήτρια, ενδεχομένω θα θέλω να πάρει το λόγο, αλλά και ο κύριος Λόμπες Αγκουιλάρ, η κυρία Μέλναρ πρώτα, η οποία είναι η σκιώδη εισηγήτρια των φιλελευθέρων. Δεν θα χρειαστώ καν το ένα λεπτό. Καταρχά θέλω να τονίσω ότι καλωσορίζουμε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά με αυτό το πρόγραμμα και εάν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να είμαστε αποτελεσματικοί τηρώντας και το των δικαιωμάτων, χρειαζόμαστε ε, ένα πακέτο για την, ε, για τα, για την προσέγγιση των δεδομένων. Δεν θα είναι ποτέ αποτελεσματική η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αν οι πολίτες δεν ε, εμπιστεύονται αυτό το σύστημα. Γι' αυτό λέω, η σημείο κλειδί είναι η προστασία των δεδομένων. Σε ό,τι αφορά τώρα το σχέδιο γνωμοδότηση, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας για τη δουλειά του. Ίσως δεν είναι τόσο τολμηρή η θέση που έχετε οι μέχρι τώρα και η γνωμοδότηση, αλλά πιστεύω ότι με τις προτάσεις που θα καταθέσουν μπορούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Τόσο ε, άτολμη η πρόταση του πάνω. Ε, ένα λεπτό μας μένει. Λόπεθ Αγιλάρ. Συγγνώμη, πρόεδρε, που ζήτησα το λόγο. Αυτή τη φορά όμως το κάνω για την κυρία Νταλή, που είναι η εισηγήτρια από τη ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και θα διαβάσω αυτό που έχει γράψει. Θέλει βέβαια να ευχαριστήσει τον εισηγήτη που έλεγε πω τόσε πολλέ από τι προτάσει τη ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών και στην Επιτροπή εδώ, αλλά και στην ακρόαση ΙΣΑ 2 που οργανώθηκε από την Επιτροπή μα. Μπορεί να είναι καλό με το νομοθέτημα, αλλά χρειάζεται να γίνουν πολλά, ιδίω ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, ε, ώστε τα διάφορα κενά που υπάρχουν να τα καλύψουμε. Και ίσω η διατύπωση θα πρέπει να αλλάξει ώστε τα δικαιώματα των πολιτών να αντικατοπτρίζονται καλύτερα και τα δικαιώματά του να γίνονται σεβαστά. υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση. Επίσης, θα έπρεπε κατά την άποψή της να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ε, προάσπιση, στην προάσπιση των δικαιωμάτων, προστασία μάλλον των προσωπικών στοιχείων, ώστε να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, να τηρούνται οι ικανός περιπροστασίας δεδομένων που θα πρέπει να καταρτιστούν γιατί Αλλιώ θα εφαρμόσουν του δικού του κανόνε ε, οι χώρε με βάση τα δεδομένα για του Ευρωπαίου πολίτε, τα οποία αποκτούν μέσω ε, κάποιες ενέργεια που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματο ΙΣΑ 2. Ολοκληρώνει λοιπόν, συντραζητώντα τη γρήγορη εφαρμογή του πακέτου μέτρων για την προστασία των δεδομένων. Όχι μόνο για την ανάγκη να έχουμε συγκεκριμένου κανόνε και ε, μέτρα για την προστασία των δεδομένων, αλλά να υπάρξει μια πραγματική κουλτούρα προστασίας δεδομένων στις υποδομές μας. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Τέλος. Συμβούλιο Κομισιόν δεν λέτε τίποτα. Όχι, δεν λέτε τίποτα. Δεν μιλάτε. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό σε καμία περίπτωση ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο η διαλειτουργικότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ που έκανα, τα έκανα τόσο βιαστικά. Και δεύτερη φορά το παθαίνετε κύριε Ελένα, να σας έχουμε βάλει στο και να σας θα στριμώ. Σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, σας πενθυμίσω, προθεσμία κατάσταση τροπολογίων 13 Μαρτίου. Η Κομισιόν με τη γλώσσα σώματος μου, μου δείχνει ή ότι θέλει να μιλήσει ή με κακολόγηψε από την πλάτη μου. Εντάξει, λοιπόν θα σας δώσω 30 δευτερόλεπτα τότε. Και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά, την καλή έκθεση. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο προηγούμενο πρόγραμμα σεβάστηκε την κοινωτική νομοθεσία και την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων σε ό,τι αφορά την ε, ε υιοθέτηση λύσεων και την, ε, το σχεδιασμό αυτών ε, λαμβάνουμε υπόσχεση σε αυτή τη διάσταση αυτή θα πρέπει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν και τους εθνικούς και του ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και πρέπει επίσης να εφαρμόζουν όλους τους νόμους που εγγυώνται την προστασία των πολιτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος πάντως θεωρώ ότι η νομοθεσία ε, περί προστασίας δεδομένων γίνεται σεβαστή ε, στη φάση προετοιμασίας ε, του προγράμματος αλλά και στη χάραξη και την υλοποίηση των λύσεων. Ευχαριστώ. I μάλιστα. Ωραία. Είπατε τα ουσιώδη. Ευχαριστούμε και την Κομισιόν. Κύριε Λένρας, έχετε κάτι να προσθέσετε. Είπα ποια είναι η προθεσμία κατάθεσης. Τίποτα άλλο. Την επόμενη φορά που θα έρθετε εδώ, θα σας βάλω πρώτο ή δεύτερο. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέλφους και το προσωπικό που εκπροσωπεί τους σκιώδης.